Carlos, are you Okay, let's start. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Συνάδελφοι, τώρα θα δούμε τα τρία πακέτα του συστήματος πληροφοριών Schengen με, τις, ε, με τα σχέδια γνωμοδοτήσεων των κυρίων Κουέλιο και Λέναρς από τον Ιούλιο και την τότε συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επί των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο που εκπροσωπεί και τον κύριο Λένος για την ανταλλαγή απόψεων. Και μετά στους και συζητητές και σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Κάρλος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις σε αυτή τη φάση. Πρώτα απ' όλα για τις τροπολογίες. Έχουμε λάβει 750 τροπολογίες για τις προτάσεις για την αστυνομική συνεργασία και το σύστημα πληροφοριών Schengen ε, και δείχνει πόση σημασία έχει για μας το σύστημα Schengen και πόσο σοβαρά το βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι. Για τη συνεργασία μα με τους Σκιώδη. Η συνεργασία μα ω τώρα υπήρξε ιδιαίτερα επικοδομητική. Έχουμε τέσσερι συναντήσει των συγκεκριτών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, Τρει πολιτικέ και μία ε, σε τεχνικό επίπεδο. Και ε, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μεγάλη πλειοψηφία για να μπορούμε να αντιμετωπιστούμε με το Συμβούλιο. Η τρίτη μου παρατήρηση για την πρόταση της Επιτροπής για το ΣΥΣ, για τις επιστροφές. Για τις επιστροφές μιλώ εκ μέρους του συναδέλφου Λένας, ο οποίος ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Για να υπάρξουν πραγματικές επιστροφές και βελτίωση του όλου συστήματος είναι σημαντικό για να υπάρξει ε, εύρυθμη λειτουργία στο σύστημα, λειτουργίας, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν και το τόνισε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, καθώς και χθες με την πρόθεση που αναφέρθηκε να ενισχυθεί η υπηρεσία των επιστροφών εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτή η βελτίωση θα βελτιώσει την ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη για τις επιστροφές καθώς και τις δυνατότητες των κρατών μελών επί του θέματος. Δεκάδε τροπολογιών υποβλήθηκαν για το θέμα αυτό. Έγινε τεχνική συνάντηση για να προετοιμάσουμε την ε, συνάντηση των σχεδόν τη επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε λίγο πολύ συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το πού θέλουμε να πάμε με την έκθεση αυτή, γιατί το σύστημα πρέπει να είναι πρακτικό. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μια ειδοποίηση σε όλε τι καταστάσει, λόγω χάρη για του επικού των χωρών που ε, βρίσκονται σε κράτηση και περιμένουν μέχρι την απομάκρυνσή τους, μέχρι να κρυθεί η υπόθεσή τους. Με τον κύριο Λέναρς θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ευθυγράμμιση. Και τέταρτη παρατήρηση για το χρονοδιάγραμμα. Τελευταία παρατήρηση για το χρονοδιάγραμμα και αφορά και τις τρεις εκθέσεις. Θέλουμε να έχουμε τελική συμφωνία με το Συμβούλιο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με αυτό κατά νου καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η θέση του Κοινοβουλίου να εγκριθεί ως τις 12 Οκτωβρίου και πρέπει να πω ότι και πάλι εδώ εκτίμησα ιδιαίτερα τις προσπάθειες των ε, σκιωδών για να πετύχουμε αυτόν τον ε, πιεστικό στόχο. Ολοκληρώνοντας, όπως έχω ξαναπεί, ε, επανειλημμένος, το ΣΥΣ είναι το μεγαλύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο και καλύτερα ε, ε, οργανωμένο σύστημα που έχουμε ως βάση δεδομένων ε, για την μετακίνηση των πολιτών και τη μετανάστευση. Ελπίζω να παραμείνει έτσι και να προσφέρουμε μεγαλύτερη επίπεδο προστασία στους πολίτες μας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να είναι εδώ η κυρία, η κυρία Μίριαν Ντάλι, η κυρία Σίπελ την αντικαθιστά. Ευχαριστώ. Δυστυχώ οι σκιώδε μα, η κυρία Ντάλη, δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ γιατί βρίσκεται στη Γενέβη, εκπροσωπώντα την ομάδα μα στι διαπραγματεύσει για την σύμβαση Μιναμάτα. Οπότε θα πω ε, κάποια λόγια εκ μέρου τη. Οι σκιώδει μα ανυπομονεί για την έναρξη των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια συμβαστική λύση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και που ε, αν όλα πάνε καλά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα εργαλεία ε, ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία αυτά είναι αναλογικά και ότι λαμβάνουν υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, όπως ανέκαθεν φροντίζαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Το ΣΥΣ είναι ένα από τα ευρύτερα, και το είπε και ο συνάδελφο Κόλλιο μόλι τώρα, ένα από τα ευρύτερα συστήματα πληροφορική παγκοσμίω και είναι και βασικό εργαλείο για την ε, κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα αυτό διευκολύνει έναν υψηλό βαθμό ε, ασφάλεια, τον ευνοεί δηλαδή, και ότι χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ιδίω τα ευαίσθητα, με υπεύθυνο τρόπο, όπω τα στοιχεία για το DNA η ομάδα μας θέλει να ε, υπογραμμίσει τέσσερα βασικά σημεία που ε, το στατούσαν σε όλες τις τροπολογίες που βάλαμε προς τον εισηγητή. Μερικές από τις παρατηρήσεις αυτές έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, οπότε δεν θα περάσω ε, στις λεπτομέρειες του κάθε μια έκθεσης και πρότασης, αλλά θα τις δω ομαδικά. Ως ομάδα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε πολλέ από τι εκφράσει και του όρου που χρησιμοποιούνται στην πρόταση αυτή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι αθώοι δεν ε, καταλήγουν ε, σοριδών στο ίδιο σημείο του συστήματος. Εδώ πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτοί που στοχεύουμε είναι οι αυτουργοί σοβαρών εγκλημάτων και ποινικών παραβάσεων και να υπάρχουν και σαφή αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι έχουν διαπραχθεί αυτά τα εγκλήματα ή αδικήματα από τους ε, εν λόγω υπόπτους. Επίσης να τονίσουμε την σημασία της αναλογικότητας. Πρέπει να διασφαλιστεί, ιδίως σε ό,τι αφορά το ποιο θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα εντό του συστήματο ΣΥΣ και για αυτό το λόγο η σκιώδη μα έχει υποβάλει σχετικέ τροπολογίε. Για την τήρηση των δεδομένων, οι σκιώδη μας έχει υποβάλει ε, επίσης τροπολογίες επί των προτάσεων, καλώντας την μείωση της πενταετούς ε, διάρκεια τήρησης των δεδομένων της Επιτροπής τα τρία χρόνια. Οι τροπολογίες αυτές επαναλαμβάνουν την ουσία των ε, αρμοδιοτήτων του επόπτη των προσωπικών δεδομένων που τα ανέφερε και στην γνωμοδότησή του για την πρόταση αυτή. Πιστεύουμε ότι βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδίω της απόφασης για την τήρηση των δεδομένων και ακόμη πιο σημαντικά της πρόσφατης απόφασης για το μετρό Επιβατών Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με αυτές τις συστάσεις. Επίσης, πρέπει να δούμε και το ε, κομμάτι της πρότασης που έχει να κάνει με τις κυρώσεις. Πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Εδώ πιστεύουμε ότι και τα κάτι μέλη και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσωπικό που έχουν πρόσβαση στο σύστημα αυτό πρέπει να βεβαιωθούν ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο λογοδοσία. Ιδίω σε ό,τι αφορά την ένταξη νέων δεδομένων στο σύστημα Schengen, την ε, κατάχρηση κάποιων δεδομένων ή την υπεξαίρεση και την ε, προσθήκη πρόσθετων πληροφοριών. Ολοκληρώνοντα, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα, αλλά είμαστε τελείω πρόθυμοι, απολύτω πρόθυμοι και αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Ντεπρέ. Σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την εργατικότητα και την προθυμία του εισηγητή μας που έχει αναλάβει όχι μόνο την ευθύνη αυτών των ντοσιέ αλλά και του άλλου που δεν είναι το δικό του. Ε, τον συγχαίρω λοιπόν για την προθυμία του και την ποιότητα των συζητήσεων που είχαμε στις συνομιλίες μεταξύ σκιωδών. Τις διοργάνωσε άριστα. Σε ό,τι αφορά Καταρχά το ΣΥΣ για τις επιστροφές. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι συμφωνώ σχεδόν με όλες τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα. Από τον εισηγητή και ιδιαίτερος οι τροπολογίες του που στοχεύουν να ενισχύσουν τις εγγύησεις στη στιγμή ανταλλαγής πληροφοριών, πρόσθετων πληροφοριών με τις τρίτες χώρες και θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα σημεία, αλλά θα εξοικονομήσω το χρόνο μας. Εγώ ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία όπου υπάρχει μια ελαφρά απόκληση στις απόψεις μας. Η δυνατότητα που προτείνει η εισηγητή στο ΣΥΣ να τηρούνται δεδομένα για τις επιστροφές επί πενταετία μετά την θέση σε ισχύ, την πραγματική θέση σε ισχύ τη απόφαση. Όταν δηλαδή κάποιο έχει ήδη φύγει το ΣΥΣ, είναι βάση δεδομένων για λειτουργικού και επιχειρησιακού σκοπούς. Δίνει συγκεκριμένε οδηγίε, μάλλον πληροφορίε για την ε, συμπεριφορά κάποιου. Ε, τη συμπεριφορά πρέπει να τηρήσει. Ε, από τη στιγμή που κάποιο έχει φύγει, δεν μα αφορά πλέον η συμπεριφορά του. Το συζήτησε ήδη με τον εισηγητή. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στο ΣΥΣ για πενταετία. Μπορεί το Eurodac να τα τηρεί. Είναι πιο χρήσιμο για τέτοιου είδου καταστάσει. Δεύτερον, ο εισηγητή προτείνει να προβλέψουμε την εισαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και όχι τα δακτυλογραφικά ε, δεδομένα όπω έχουν ονομαστεί. Νομίζω ότι καλά το προτείνει μεν, αλλά από την άλλη όσο πιο πολλέ πληροφορίε υπάρχουν τόσο, το τόσο καλύτερα. Έτσι λοιπόν δεν θα επιφυλαχθώ να υποβάλω σχετικέ τροπολογίε για το τι ε, πληροφορίε μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε στο σύστημα. Για τη συνεργασία τώρα των συνοροφυλακών με τι αστυνομικέ δυνάμει. Συμφωνώ κατά πολύ με τι προτάσει του εισηγητή. Συμμερίζομαι τι αμφιβολίε του για την υποχρέωση κάθε κράτου μέλου να διαθέτει ε, εθνικό αντίτυπο, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να μην υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν εθνικό αντίτυπο, αλλά να ενισχύσουμε απλώς την δομή του κεντρικού συστήματος, κατά τρόπον ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα ε, με περισσότερο αποτέλεσμα, με περισσότερη ε, αποδοτικότητα. Επίσης, ο εισηγητής σωστά εντοπίζει ότι πρέπει κάποια αιτήματα πληροφόρησης να γίνονται δεκτά. Το κείμενο α, ε, ορίζει ότι μετά από αίτημα για πληροφορίες προς των πληροφοριών από κάποιον συνοριοφύλακα ή αστυνομικό, το γραφείο ΣΥΡΕΝ απαντά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε μια μέγιστη προθεσμία 12 ωρών. Όμως έχουμε ε, οργανώσει ε, γραφεία που πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα για τα θέματα της τρομοκρατίας, του εντοπισμού τρομοκρατών και εκεί είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος που τρέχει. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε στη διορία το διάστημα των 12 ωρών που προτείνει ο κύριος Χαίλιο. Θα πρέπει τα γραφεία ΣΥΡΕΝ να απαντούν αμέσως, ε, το δυνατόν πιο γρήγορα εφόσον αυτό το κάνουν για την ε, τρομοκρατία. Επίσης, η η ιδέα ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τρομοκρατία πρέπει να κοινοποιούνται στη Europol. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να δούμε τι εννοώ. Ας πούμε ότι έχει γίνει μια επίθεση στη Γερμανία. Ότι η γερμανική αστυνομία εντοπίζει ε, το όνομα έστω του υπόπτου. Αλλά δεν, έχει χρόνο να το εισάγει, δεν είχε το χρόνο να το εισάγει στο ΣΥΣ. Και αυτός ο δράστης έχει φύγει από τη γερμανική επικράτεια και έχει πάει στο Βέλγιο ας πούμε και έχει εντοπιστεί στο Βέλγιο γιατί το έχει σημάνει η Γαλλία. Οι μόνες χώρες που ξέρουν ότι είναι ε, στο Βέλγιο και μπορεί να πάρει πτήση για να φύγει είναι η Γαλλία και το Βέλγιο σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να σκεφτούμε αν συστηματικά πρέπει να το ε, μαθαίνει αυτομάτως η Europol και αν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι επιχειρησιακή ανάγκη, πιστεύω, γιατί αλλιώ θα υπάρχουν τριγωνικά ελλείψει στο σύστημά μα και θα πρέπει να δούμε πώ θα λειτουργήσουν τα δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ε, αυτά είναι μερικά από όσα θέλω να εντοπίσω και να υπογραμμίσω. Θα τα συζητήσω ξανά με τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ για την υποκοδομητική ατμόσφαιρα και προσβλέπουμε στι επόμενε συνομιλίε μα. Ευχαριστούμε. Τώρα, η Μαρίν Κριστίν Βερζιά έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη γιατί δεν έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το κείμενο, σας το είπα ήδη. Δουλεύω όμως το σύστημα εισόδων-εξόδων και μου είναι δύσκολο όλα αυτά να τα βάλω σε μια γενικότερη λογική, η οποία έτσι καλλιώς με ανησυχεί. Κυρίως, θα έλεγα, του τρίτου κειμένου ΣΥΣ, αυτό που ονομάζουμε ΣΥΣ επιστροφών. Γιατί πίσω από το κείμενο αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην τρομοκρατία και την εγκληματικότητα από τη μια και την παράτυπη μετανάστευση από την άλλη. Κάτι το οποίο μου είναι δύσκολο να δεχτώ, ακόμα και αν αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέμε για την προστασία, τον έλεγχο των συνόρων κτλ. Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη μεριά είναι εντύπωση που μένει και αυτή μου δημιουργεί πρόβλημα και εξαρτάται τελικά από τις αρχές εκείνες οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι σε θέση να μπορώ να έχω μια γενική λογική μέσα στην οποία να γράφω όλα αυτά. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η νομοθεσία των χωρών μελών δεν είναι εναρμονισμένη όσον αφορά το θέμα έτσι κι αλλιώς της ε, νόμιμης μετανάστευσης, της κανονικής μετανάστευσης ούτε καν για το θέμα των προσφύγων. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τα συστήματα αυτά με τα οποία θα στέλνονται σήματα πώς θα λειτουργήσουν όταν πρόκειται για κάποιον που ζητάει άσυλο. Οι εξελίξεις είναι ανησυχητικέ. Έχουν ε, απελαθεί άνθρωποι από τις χώρες μας. Βέλγιο, για παράδειγμα οι βελγικές αρχές με τις αρχές του Σουδάν συνεργάζονται για να εντοπίσουν ανθρώπους και να ευνοήσουν έτσι τις επιστροφές. Αν λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα στην Ευρώπη με συστηματικά σήματα που θα στέλνονται, ανησυχώ για το τι θα γίνει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα προχωρήσουν οι αξίες της. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια αρχή που ισχύει τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και για τους πολίτες τρίτων χωρών. Επιμείναμε για τις τροπολογίες, δεν μιλάω μόνο για τις τροπολογίες εδώ επί της αρχής, τις οποίες ε, έχουμε υποβάλει, αλλά επιπλέον θέλουμε και μια επικοδομητική προσέγγιση, ώστε το σύστημα αυτό, αν μη τι άλλο, να σέβεται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές που στηρίζει ότι έχει. Γι' αυτό λοιπόν και θα έχουμε τροπολογίες οι οποίες θα αναφέρονται ακριβώς σε αυτά και στο θέμα της αναλογικότητας σε σχέση με το στόχο μας. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σας και στο παρελθόν και ξέρω ότι σας νοιάζει αυτό. Ο κάθε τελικός μας στόχος δεν εξυπηρετείται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε το θέμα της κοινωνικής ε, εικόνας κλπ. Και η επαλήθευση επίσης των δεδομένων. Διότι τελικά θα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν όλα αυτά στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας. Τώρα το δικαίωμα προσφυγής των ενδιαφερόμενων κυρίως όταν πρόκειται για ανθρώπους από τρίτες χώρες και μάλιστα όταν δεν είναι τακτοποιημένη η κατάστασή τους, είναι παράτυπη δηλαδή, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα και τροποποίησή τους άπαξ και είναι εσφαλμένα, ακόμα και αποστεριόρι αν το δικαίωμά τους σε εγκατάσταση. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν όλες εγγυήσει οι οποίες συνοδεύουν την προστασία δεδομένων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις θέσεις μας για αυτά τα ζητήματα και κυρίως για την τήρηση και το σεβασμό της σύμβασης της Γενέβης που πάει όλο και χειρότερα. Γιατί οι χώρες μέλη δεν την εφαρμόζουν καλά. θα έπρεπε να βάζουμε ρήτρε ασφάλειας σε αυτά που εφαρμόζουν οι χώρες μέλη και όχι να ξεχνάμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σύμβαση της Γενέβης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδες εισηγητές εδώ που να ζητούν το λόγο. Η κυρία Τσινίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους που εργάζονται επί του θέματος αυτού τον κανονισμό για το σύστημα ΣΥΣ. Εξαιρετική η δουλειά τους, διότι πρόκειται πραγματικά για ένα κείμενο πολύ περίπλοκο. Θέλει να ρυθμίσει ένα εργαλείο που θεωρώ καθοριστική σημασία για την ασφάλεια, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να σεβεται τα δικαιώματα των πολιτών, όπω μόλι υπογραμμίστηκε από τον εισηγητή στην παρέμβασή του. Ήθελα εδώ να σταθώ σε μια συγκεκριμένη πτυχή. Το γεγονός ότι το σύστημα ΣΥΣ είναι αναγκαίο κατά την άποψή μου για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την ε, εξαφάνιση ανηλίκων. Εδώ μαζί με την ε, οριζόντια ομάδα για τα δικαιώματα των ανηλίκων και μετά από δικές τους συστάσεις υπέβαλα κάποιες τροπολογίες. Ε, καλύτερα συμφέροντα των ανηλίκων πρέπει πάντοτε να την υπόψη κατά την εφαρμογή του συστήματο. Ε, αυτό ισχύει για τις τροπολογίες που στόχο έχουν να βεβαιώσουν ότι οι σημάνσεις που αφορούν ανηλίκους γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με αρχέ που είναι υπεύθυνε για την προστασία των ανηλίκων. Ιδίω στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων και που θεωρούνται εξαφανισμένοι, είναι σημαντικό η συλλογή δεδομένων, η τήρηση και η πρόσβαση σε αυτά να έχουν πάντοτε σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία του ανηλίκου. Επίσης, μια άλλη πτυχή, όπως διακομματική ομάδα θελήσαμε να πάρουμε θέση με κάποιε τροπολογίε, έχει να κάνει ακριβώ με τη διαφορετική θέση των ε, υποεξαφάνιση ανηλίκων. Εκεί πρέπει να ε, εξεύρουμε ένα μέτρο εξειδικευμένο, το οποίο να λειτουργεί ανάλογα με την κατάσταση, τις συνθήκε του κάθε ανηλίκου και οι αρμόδιοι να μπορούν να μεταβάλουν την απόκρισή τους ανάλογα με το τι συμβαίνει. Ένας αλλοδαπός ανήλικος, ασυνόδευτος που φτάνει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και μετακινούμενος ε, ξαφανίζεται, χάνουμε τα ίχνη του, είναι πολύ διαφορετικός από ένα παιδί που είναι θύμα διεθνούς απαγωγής, λόγου χάρη. Εάν δεν δοθούν λοιπόν διαφορετικές αποκρίσεις στις διαφορετικές περιπτώσεις των παιδιών, δεν υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις διάφορες συνθήκες, ε, δεν θα είναι αποτελεσματική παρέμβασή μας ε, στις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε ακριβώς με παιδιά αυτό θελήσαμε να τονίσουμε με τις τροπολογίες που υποβάλαμε, την υποχρέωση πάντοτε οι συγκεκριμένες αρχές με αρμοδιότητες για την προστασία των ανηλίκων να παίρνουν πάντοτε μέρος στην ε, αποτίμηση των διάφορων υποθέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε περίπτωση τον συνάδελφο για την πολύ καλή του δουλειά, αλλά είμαι βεβαίω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για το κείμενο αυτό για να φτάσουμε σε μια λύση συνενετική. Πρόκειται για ένα εργαλείο καθοριστικό για την αστυνομική και συνεργασία και καθοριστικό για την προστασία των δικαιωμάτων και όπως ε, υπενήχθηκα προηγουμένως, όλος ιδιαίτερος για την προστασία των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων που είναι τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από το δίποτα άλλο, επενθυμίζω ότι η δικιά μου πολιτική ομάδα είναι κατά τη συμφωνία Σέγγελ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχει η συμφωνία αυτή τόσα χρόνια. Ε, τουλάχιστον να προσπαθούμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματική για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Και αυτό και κάνει πρόταση κανονισμού. Είναι μια πρόταση που θέλει να χρησιμοποιείται το σύστημα πληροφοριών Schengen προκειμένου όσο γίνεται καλύτερα να βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια όσοι παράνομα βρίσκονται μέσα σε αυτή. Υπάρχουν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Κάποιες ενισχύουν αυτό το στόχο, οπότε πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτές. Τρία παραδείγματα θα σας δώσω. Τροπολογία αριθμός 5, η οποία επιτρέπει για 5 χρόνια να κρατάμε τα στοιχεία όσον αφορά τους ε, ανθρώπους ε, για τους, οι οποίοι δεν έχουν φύγει από τη χώρα. Υπάρχει αυτό η οποία αναφέρεται ε, επίσης στη σήμανση των ατόμων αυτών και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα που είναι η αριθμός 20 η οποία προτείνει στην έκταση της σχετικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας να αναφέρονται τα στατιστικά δεδομένα. Να λοιπόν κάποιες τροπολογίες που δείχνουν πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό Σέγγεν για να αποφύγουμε αυτήν την ε, ανατροπή που μας φέρνει η μετανάστευση. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε, λέει ο Η μεταναστευτική κρίση και εκείνη της προστασίας μας δοκιμάζει τα συστήματα ασφάλειας και τα συστήματα πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά πρέπει να εξυπηρετούν τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Τα νέα μέτρα και οι νέες διατάξεις έχουν ως στόχο ακριβώς να διασφαλίσουν καλύτερη προστασία στα ευρωπαϊκά σύνορα. Σας Παρακαλώ λοιπόν να στηρίξετε τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τα άτομα τα οποία επιστρέφονται, ακόμα και αν δεν υπάρχει απαγόρευση επιστροφής. Οι αρχές δηλαδή θα μπορούσαν έτσι να έχουν μια ιδέα του κινδύνου για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιστρέφονται. Το σύστημα, οπότε, στη συνέχεια θα μπορούσε να χρησιμοποιείται καλύτερα και όντως να διασφαλίζει την προστασία. Και μια που μιλάμε για ασφάλεια, η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία 100% υλοποιεί όλα τα μέτρα Πρέπει να μπει λοιπόν στο χώρο Σέγγεν και είναι αυτή η έκκληση που κάνω προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει ότι πραγματικά δίνει σημασία στην ασφάλεια στα σύνορα και την προστασία τους. Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στον κύριο Έκατ Μπαρίτσα. εκ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ναι, από πλευράς της Προεδρίας μπορώ να σας ενημερώσω κάπως για τους ε, φακέλους αυτούς όσο μπορώ περισσότερο. Αυτή την εποχή κλείνουμε τις διαδικασίες για τους φακέλους αυτούς και είναι καλό που ακούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Συμβούλιο προχωράμε με το ίδιο χρονοδιάγραμμα λίγο πολύ προσπαθούμε να έχουμε την ε, γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο συγχρόνως με την ψηφοφορία που θα έχει το Κοινοβούλιο. Άρα μπορούμε μετά όσο γίνεται πιο γρήγορα να αρχίσουμε το τριμερή διάλογο. Θέλουμε και εμείς να έχουμε τη συμφωνία πριν από τα τέλη της χρονιάς, όπως είπε και το Κοινοβούλιο σήμερα ότι θέλει. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε τον ίδιο βηματισμό και τα όσα άκουσα σήμερα με κάνουν να πιστεύω ότι ο στόχος είναι κοινός μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θέλουν να έχουμε στη διάθεσή μας το καλύτερο σύστημα που να εφαρμόζεται και όσο γίνεται καλύτερα ώστε να εξυπηρετούνται όλοι και να διασφαλίζεται και η προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την Επιτροπή τώρα. Η κυρία Έρκα Γιάντσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Λίβερ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι σχόλια μετά από πολλή σκέψη και δείχνει ότι είσαστε και ειδικοί στο θέμα. Κυρίως τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκαν και στο Συμβούλιο. Και βλέπω ότι αυτό που ενδιαφέρει τις χώρες μέλη και αυτό που ενδιαφέρει εσάς είναι το ίδιο. Στη... Αυτά που συζητήθηκα στο Συμβούλιο αντικατοπτρίζονται και στις δικές σας συζητήσεις. Γι' αυτό και προσβλέπω σε μια εύκολη συμφωνία μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τη Europol. Και ευχαριστώ τον κύριο Ντεπρέ για αυτά που είπε. Γιατί αρχίζει να χρησιμοποιεί ενεργά το σύστημα Europol. Έχει ήδη χρησιμοποιήσει πολύ το σύστημα αυτό με μια απλή τεχνική παρέμβαση. Και ήδη λέμε στην πρότασή μας ότι θα συνδεθεί η Europol με συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε πραγματικό χρόνο θα έχουν λοιπόν κοινοποίησει για το κάθε σήμα που θα στέλνετε. Είναι συνεπώς ένας πολύ καλός τρόπος να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με την Europol και να συμμετέχει άρα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Εδώ έχουμε προχωρήσει λοιπόν πολύ καλά. Θέλω όμως επίσης να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τις προδιαγραφές που ήδη προβλέπονται στην υλοποίηση του νομικού μέσου. Είπατε ότι αποτελεί κλειδί για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο από την τρομοκρατία, αλλά και από το έγκλημα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Αν νιώθουν ότι είναι προστατευμένοι και ότι ο περίγυρός τους είναι ασφαλής και δεν κινδυνεύουν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις ίδιες προδιαγραφές και να μην τις μειώσουμε. Η τροπολογία σας αναφέρεται στο άρθρο 36. Εγώ όμως εδώ θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στο μέλλον για παντό είδου έγκλημα και όχι μόνο για την τρομοκρατία. Για οποιοδήποτε έγκλημα δηλαδή όπου προβλέπεται μία ποινή πάνω από τρία χρόνια. Γιατί μέχρι τώρα όταν είναι κάτω από τρία χρόνια οι αρχές δεν ε, κάνουν όλα αυτά. Επίσης, ταραχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όπω και η τρομοκρατία και στους μαγαζάτορες. Στη Γερμανία το είδαμε αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην ασχολούμαστε μόνο με την τρομοκρατία αλλά και με άλλου είδους εγκλήματα και με περιπτώσεις δηλαδή όπου το επίπεδο ποινής είναι χαμηλό. Τώρα για τη διατήρηση των δεδομένων. Είπατε ότι προτιμάτε να κρατήσετε την τρέχουσα περίοδο. Όταν μιλάμε για διατήρηση, δεν είναι ο πιο σωστός όρος. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να διατηρούνται όσο εξακολουθούν να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο συλλαμβάνεται ή κάποιος αγνοούμενος βρεθεί Εγώ δεν θα μιλούσα για διατήρηση, θα μιλούσα για αναθεώρηση, δηλαδή μια περίοδο μετά από την οποία μπορούν να αναθεωρηθούν τα δεδομένα. Και για να μην έχουν όλο το άκθος οι αρχές, πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να κρατήσουμε την πενταετή περίοδο. Και όταν ο στόχος έχει επιτευχθεί, τότε μπορούν να διαγράφονται. Και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες για γνωούμενους για ευάλωτα άτομα, ίσως θα έπρεπε να είναι ένας χρόνος. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κίνδυνος από το να έχουμε μια μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης ή μάλλον αναθεώρησης. Όσον αφορά τις επιστροφές, είπατε ότι είναι προτιμότερο να έχουμε τα πέντε χρόνια διατήρηση των δεδομένων εγώ θέλω εδώ να τονίσω ότι όπως είπε και ο κύριος Ντεπρέ, είναι ένα σύστημα όπου τα διάφορα σήματα είναι για τις αρχές και τους βοηθούν να αποφασίσουν τι δράση πρέπει να πάρουν. Δεν είναι μόνο προς ενημέρωση. Εδώ μπορεί να τίθεται θέμα προστασίας δεδομένων για το υποκείμενο των δεδομένων. Πάντως για το στόχο των επιστροφών και τις αποφάσεις, τα δεδομένα δεν πρέπει να είναι στο ΣΥΣ, αλλά στο Eurodac ή κάπου αλλού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. για τα υποχρεωτικά αντίγραφα των χωρών Μιλάμε για αλφανομερικά δεδομένα στο κεντρικό σύστημα. Τεχνικά μιλώντας, αποτελείται όμως το σύστημα αυτό από διαφορετικά στοιχεία από δίκτυα και τα δίκτυα αποτελούνται από πολλά στοιχεία επίσης. Και δυστυχώς ε, προχωράει η αλυσίδα των στοιχείων αυτών για την ε, προστασία των ε, ανθρώπων πρέπει να υπάρχει ένα backup, ένα αντίγραφο. Και ξαναλέω ότι το εθνικό αντίγραφο υποβάλλεται σε πολύ αυστηρές προδιαγραφές προστασίας και συνέπειας. Το αντίγραφο στο κεντρικό σύστημα περνάει από ελέγχου τακτικά. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου διαφορά. Είναι μηδενική αυτή η διαφορά. Φάνηκε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε το εθνικό αντίγραφο. Ακόμα και αν το δίκτυο δεν ήταν διαθέσιμο, η χώρα μέλος μπορούσε να προχωρήσει το έργο της. Γι' αυτό θα ήθελα να διατηρηθεί αυτό στην πρόταση. Προσβλέπουμε σε διάλογο μαζί σας και στις συζητήσεις που θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε και με τα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας βοήθησαν πολύ. Επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποια σχόλια. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τις πολιτικές τους ομάδες για τα σχόλιά τους. Στρέφομαι προς την κυρία Σίπελ και θέλω να της πω ότι μοιραζόμαστε τις ανησυχίες που έχει, τις ημεριζόμαστε για την πρόσβαση και για τις κυρώσεις κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και το ίδιο συνισχύει και με τους σοσιαλιστές. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια, από την ίδια πλευρά. Τώρα ως προς τα σχόλια του κυρίου Ντεπρέ. Θα ήθελα να πω ότι τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ γιατί ε, συμφωνούμε για τα εθνικά αντίγραφα για το γεγονός ότι στόχος τους είναι να ενισχύσουν την σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του κεντρικού συστήματος. Και ευχαριστώ και την ομάδα των φιλελεύθερων γιατί κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Συμφωνώ και με το σχόλιο σας κύριε Ντεπρέ όταν αναφερθήκατε στην ανάγκη εξασφάλισης μιας πιο αποτελεσματικής απάντησης από το σύστημα ΣΥΡΕΝΕ. 12 ώρες είναι υπερβολικά πολλές όταν έχουμε πραγματικά ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης, άμεσης απάντησης, κυρίως ε, σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά όχι μόνο. Έρχομαι τώρα ε, στην κυρία Βεχουσιά και στα σχόλιά της για να πω ότι συμμερίζομαι τα σχόλιά σας κυρία Βεχουσιά Πράγματι, δεν θέλουμε να υπάρξει σύγχυση μεταξύ τρομοκρατίας, μεταναστευτικών ροών και προσφύγων. Συμφωνώ απολύτω και ό,τι μπορεί να γίνει για να αποφευθεί αυτή η σύγχυση θα το κάνουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι για όλους και όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Συμφωνώ απολύτως και συγχαίρω και ευχαριστώ την κυρία Βερσία για την τροπολογία της για τα δικαιώματα των υπηκών τρίτων χωρών εντός συστήματος και πιστεύω ότι είναι κάτι που πραγματικά μπορούμε να προσθέσουμε στην τελική έκθεση. Αν μου επιτρέπει όμως η κυρία Βερσιά, θα ήθελα ε, να πω, θα τολμούσα να πω ότι για την ΚΟΕ, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο εύκολο να έχουμε μία σωστή έγκριση με το υφιστάμενο σύστημα, με τις αρμοδιότητες και τον έλεγχο της διατήρησης ε, και των αντιγράφων, παρά το νέο σύστημα. Καταλαβαίνω δηλαδή το σκεπτικισμό της κυρίας Βεχσιά για το νέο σύστημα που αναγγέλλεται και τις επιφυλάξεις της. Όμως, πάνω σε κάτι που ήδη έχουμε, που λειτουργεί καλά, που ήδη ξέρουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, νομίζω ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε το σύστημα που έχουμε, το υφιστάμενο. Για την κυρία Κινίτσι. Ε, είμαστε στο ίδιο μήκο Πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν είναι ένα από τα... Έχει, παρουσιάζει το εξή ενδιαφέρον. Ενισχύονται οι εγγυησει, οι για τους ανηλίκους, για τα παιδιά, και εγώ αλλά και άλλες δύο πολιτικές ομάδες έχουμε προτάσεις για να το εγγυθούμε αυτό ε, επισημάσεις ε, και να σημαίνει ειδικό συνέγερμος νωρίτερα για τα παιδιά, για τους ανηλίκους διατάξεις προστασίας των ανηλίκων και ποτέ δεν ξέχασα αυτά που μας είπε η Europol για τα 10.000 εξαφανισμένα παιδιά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όνειδος για εμάς και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον δεν θα, ε, θα αποφύγουμε. Εν πάση ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ για, τα, για τη βοήθειά σας. Ο κύριος Λεμπρετών ε, σχολίασε τα σχόλια του κύριου Λεμέρ, θα τα διαβιβάσω στο συνάδελφο και ο κύριος Ράντεφ το ίδιο. Τα σχόλιά του τα Απίστηνε κυρίως στο θέμα των επιστροφών. Όμως ο κύριος Ράντεφ ε, είπε κάτι για τη Βουλγαρία και θέλω να το προσυπογράψω. Ε, να μην ξεχνάμε ότι ήμουν ειδικό εισηγητής για τη διεύρυνση του χώρου Σέγγεν και τη συμπερίληψη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν η επαλήθευση ε, του γεγονότος ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και καταλήξαμε στο συμπεράσμα στο Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και στο Συμβούλιο με ομοφωνία ότι έχουν επαληθευτεί όλα τα συμπεράσματα, αλλά δεν υπάρχει κανένας ούτε πολιτικός ούτε τεχνικός λόγος που μπορεί να εμποδίσει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα σχόλια θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά τους. Είμαι αισιόδοξο, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Ελπίζω λοιπόν μέχρι τα τέλη της χρονιάς σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ για την απίστευτη δουλειά σας, πάρα πολύ επαγγελματική, Κάρλος. Ψηφοφορία θα έχουμε στις 11 και 12 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η νομιμοποίηση παράνομων προσόδων και εσόδων μέσω της, ε, του ποινικού δικαίου Εισηγητής είναι ο κύριος Κοράο. Είχαμε μία αρχική παρουσίαση στις 29 Ιουνίου του 2017 στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η προτινόμενη οδηγία παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2016 και βασίζεται στη σύμβαση του 2005 του, Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την αναζήτηση, την ανείχνευση, την δέσμευση και την δίμευση των προσόδων του εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα. Και βασίζεται και στις συστάσεις FATF, δηλαδή στην ε, Task Force, την ειδική ομάδα για την χρηματοοικονομική δράση, Financial Action Task Force. Όμως αυτή η πρόταση οδηγίας υπερβαίνει αυτά τα δύο νομοθετικά οργαλεία. Έχουμε Έχουμε τον αριθμό αυτών των αδικημάτων, το self-laundering, την αποσύνδεση ε, των αδικημάτων που έχουν να κάνουν με το ξέπλυμα χρήματος από την πεποίθηση ε, σύμφωνα με την οποία η ποινική δραστηριότητα δημιούργησε αυτή την ιδιότητα, αυτή την ιδιοκτησία. Και υπάρχει και το θέμα της έξω εδαφικότητας. Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο υιοθέτησε τη γενική του προσέγγιση στις 8 Ιουνίου του 2017. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κοράο, τον εισηγητή. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους Κιώδης για την στάση τους, τη συνεργασία που είχαμε και για τη δουλειά μας τους τελευταίους μήνες. Δουλειά προπαρασκευής, συζήτησης, συνομιλιών για να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο σαφές να έχουμε ένα κείμενο, γιατί η οδηγία αυτή κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική, ξεκάθαρο. Μιλάμε για ένα εναρμόνιση επιχειρησιακών συστημάτων, συστημάτων ε, της νομοποίησης εσόδων, ενό εγκλήματο απεχθού που προκύπτει και έχει να κάνει με τις ομάδε οργανωμένων εγκλήματο, με παράνομε δραστηριότητε. Ε, υπάρχει ολόκληρος ε, μηχανισμός ανταγωνισμού μέσα στην ε, νόμιμη αγορά για να προλάβουν όλοι αυτοί να νομιμοποιήσουν και θα πρέπει να δώσουμε στις αρχές μας, στις δικαστικές αρχές, τους δικαστές, τη δυνατότητα να τιμωρήσουν αυτές τις πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν η οδηγία αυτή να είναι αυτό το βήμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τιμωρήσουν αυτό το απεχθές έγκλημα. Θα ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη. Η πρότασή τη είναι μια καλή πρόταση οδηγία. Επί τη οδηγία αυτή μπορέσαμε να ε, εργαστούμε και ήταν ένα πολύ καλό σημείο αφετηρία. Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλήρε κείμενο και ξεκάθαρο. Γι' αυτό θα σταθώ στα πιο ακαθόδη σημεία, αυτά που ήταν δυσκολότερο να εξηγήσουμε στο κείμενο, αλλά καταφέραμε με 27 τροπολογίες που αφορούν διαφορετικά σημεία να βελτιώσουμε κάπως την πρόταση της Επιτροπής. Τα βασικά σημεία αφορούν τον ορισμό ακριβό του αδικήματος της ε, νομιμοποίησης εσόδων, που είναι σίγουρα ένα, μια ενέργεια με δόλο, ε, και θα πρέπει να ορίζεται αν υπάρχει συγκεκριμένος βόλος για να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το βάρος της απόδειξης. Σε ό,τι αφορά την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, ένα ε, εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην Ιταλία λόγω χάρη για να τιμωρήσουμε, για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και να δώσουμε στους δικαστές ένα εργαλείο, συγκεκριμένο εργαλείο, για να πλήξουν το οργανωμένο έγκλημα στα περιουσιακά του στοιχεία. Ε, εδώ ε, η κλασική φράση ήταν ακολούθα τα λεφτά και θα βρεις τα, ε, την εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό το έλεγαν ο Φαλκόνε και ο συνεργάτης του. Εδώ πρέπει να δούμε τη δίμευση και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικέ ε, δραστηριότητε. Ένα άρθρο πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε συμπεριλάβει την αντιστροφή του βάρου τη απόδειξη ε, με ξεκάθαρο τρόπο. Υπάρχει κατάσχεση και αφήνουμε ε, μια σχετική ισορροπία για να μπορεί και ο κατηγορούμενος να διασφαλίζει τα δικαιώματά του ο δικαστής μπορεί να ακολουθήσει επιχειρηματολογία βάσει της κατάσχεσης και υπάρχει και η δυνατότητα της ελεύθερης άσκησης, ε, της ελεύθερης πυθούς με μια επιχειρηματολογία. Επίσης, η εγκληματική δραστηριότητα και τα προϊόντα της εγκληματικής δράσης. Υπάρχει ένας, ένα, μια διπλή πορεία για, την, ε, για τον εντοπισμό των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έχουμε δύο εξαιρέσεις για, για το διπλό τεκμήριο εγκληματικής δράσης και οι δύο εξαιρέσει είναι ακριβώς μια σειρά από αδικήματα που θεωρούνται σοβαρά, όπως η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία ή η διαφθορά, ενώ η δεύτερη εξαίρεση είναι οι χώρες υψηλού κινδύνου όπως τις έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης έχουμε προβλέψει συγκεκριμένε κυρώσεις, τις οποίους θεωρούμε τις οποιες θεωρουμε δραστικες και αποτρεπτικές, όπως η μόνιμη υπαγόρευση να έχει κανείς οποιαδήποτε συμβασική σχέση με τις δημόσιες αρχές. Βεβαίως, ε, εργαστήκαμε με ένα, ε, σε ένα πολύ καλό κλίμα με τους ε, σκιώδεις και θα κοιτάξουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές τροπολογίες μετά από τις επόμενες συνομιλίες μας για να έχουμε μια ισχυρή θέση ως Κοινοβούλιο τη δημοτεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε να καταλήξουμε σε αίσιο πέρας στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, στις 12 Οκτωβρίου προβλέπεται η παρουσίαση των τροπολογιών εδώ στην Επιτροπή μας, ως προς το χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Θα παρουσιαστούν στις 19 Οκτωβρίου, στις 13 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και ελπίδα μου είναι να πετύχουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια ως τον Νοέμβριο για να ολοκληρωθεί το ντοσχέ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μια δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Η Μόνικα Χολμάγερ, που είναι η σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά και τους υπόλοιπους σκιώδης εισηγητές για την εξαιρετική τους συνεργασία προβήκαμε σε έντονες ανταλλαγές απόψεων και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση του, η οποία είναι μια πολύ καλή βάση για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ε, λαμβάνει κάποιος χρήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει εάν είναι νόμιμο εντό αγωγικών, εάν μπορεί να τα δεχτεί ή εάν υπάρχει ενδεχόμενο να προέρχεται αυτό το χρήμα από ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να το δηλώσει. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο, υπάρχουν συγκεκριμένα δικήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά. Και τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένο όριο χρηματικό ή συγκεκριμένα δικήματα Για μένα όλα αυτά είναι πολύ καλές ιδέες. Εάν θέλουμε να περιορίσουμε το κείμενο στην τρομοκρατία και στο λαθρεμπόριο όπλων, αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται. Ή αν θέλουμε να διευρύνουμε το κείμενο για να περιλάβει και την φυσικά παράνομη δραστηριότητα του λαθροπορείου ανθρωπίνων οργάνων ή της εκμετάλλευσης ανηλίκων. Όλα αυτά οφείλουμε να τα έχουμε υπόψη μας. Ίσως είναι προβληματικό να αναφέρουμε επιγραμματικά δύο περιπτώσεις και να αποκλείουμε όλες τις άλλες από την ρητή αναφορά. Αξίζει να συζητηθεί νομίζω αυτό. Η κυρία Γκόμες ε, ασχολήθηκε πολύ με ένα θέμα και είναι πολύ θετικό και αναφέρομαι στις ε, εταιρείε ε, βιτρίνα, τις εταιρείε ουσιαστικά που έχουν μόνο μία ταχυδρομική θηρίδα χωρίς γραφεία. Και μετά αναφέρομαι επίσης και στα μικρά εμβάσματα, πολλά μικρά εμβάσματα τα οποία θρηστικά καταλήγουν στο να διοχετεύσουν από το ένα σημείο στο άλλο τεράστια ποσά κάποιοι είναι εξαιρετικά ισχυροί και επινοητικοί ε, στην προσπάθειά τους να περιπλέξουν τα πράγματα για τις ενδιαφερόμενες αρχές. Τώρα, ως προς την ε, δέσμευση και τη δίμευση των περιουσιακών στοιχείων, νομίζω ότι ήδη υπάρχει σχετική οδηγία. Θα την ε, αναφέρουμε συγκεκριμένα, θα βάλουμε συγκεκριμένη παραπομπή ή όχι. Αυτό ίσως θα ήταν κάπως προβληματικό. στο κείμενο πράγματι θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτή την οδηγία που υπάρχει ήδη. Να αποφύγουμε όμως τις επικαλύψεις και τους ε, πλεονασμούς. Κάποια ζητήματα μπορούμε ήδη να τα διευκρινίσουμε μεταξύ μας εδώ σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε. Νομίζω ότι στις διαπραγματεύσεις θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια από κοινού λύση. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω, η κυρία Γκόμες, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοράο για την έκθεσή του, για τις συναντήσεις με, με τους εμπειρογνωμόνες που ε, οργάνωσε, εξαιρετικά χρήσιμες συναντήσεις για εμάς και για τις δημιουργικές ιδέες θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοράο είχε πολλές ε, δημιουργικές ιδέες και τις υπεριέλαβε στην πρόταση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό, εξαιρετικά σημαντικό. Με την Επιτροπή για τα Panama Papers καταλήξαμε σε συγκεκριμένα ευρήματα και πρέπει να αντλήσουμε από αυτά τα διδάγματα για να κάνουμε τώρα καλή δουλειά. Είναι μια ε, εξαιρετική ευκαιρία αυτή που μας παρουσιάζεται έτσι ώστε ιδιοκτικές και δικαστικές αρχές καθώς και οι αρχές επιβολής του νόμου, οι εισαγγελικέ αρχές γενικότερα να έχουν αποτελεσματικά εργαλεία, να έχουν εργαλεία που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όταν προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτού του είδους την παραβατικότητα και υπενθυμίζω ότι μιλούμε εδώ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αυτό το στοιχείο συχνά διαφεύγει της ε, προσοχής ενός κράτους μέλους όταν εξετάζει το δικό του νομικό πλαίσιο ο καθένας. Όμως, εμείς ως μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουμε αυτό το θέμα να το έχουμε στο προσκήνιο. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν αποτελεσματικά να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, ε, θα πρέπει αποτελεσματικά να καταπολεμήσουν την χρηματοδότησή της. Και θα πρέπει να γίνουν πολλά γιατί ήδη οι εγκληματικές οργανώσεις αξιοποιούν όλα τα παραθυράκια των χρηματοπιστωτικών συστημάτων αλλά και των φορολογικών συστημάτων των χωρών μελών για να προωθήσουν τις παράνομες επιδιώξεις τους. Πιστεύω λοιπόν ότι στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία με τον αρχών επιβολής του νόμου, διοκτικών αρχών και εισαγγελικών, και θα ήθελα να τονίσω σε πόσο, σημαντικό είναι το στάδιο στο οποίο είμαστε τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη δίωξη και την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος μόνο όταν υπάρχει καταδίκη για... για τεκμηριωμένο αδίκημα ή τεκμήριο αδικήματος predicate offense. Έχουμε την αρχή του follow the money. Ακολούθησε το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το έχουν επισημάνει ε, ε επανειλημμένως οι διοκτικές αρχές. Όπως είπε και η Μόνικα Χολμάιερ, Υπάρχει κάτι που μπορεί να επιτευχθεί εάν υπάρξει απευθείας παραπομπή στην οδηγία που αναφέρεται στην δέσμευση και ενδεχομένω κατάσχεση ή δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Με αυτή την αναφορά μπορούμε να ενισχύσουμε ε, τη διατυπώση. Και θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό που προτείνει ο κύριος Κοράο όταν μιλά για εγκληματική δραστηριότητα που ε, δημιουργεί περιουσιακά στοιχεία και λαμβάνει χώρα στην επικράτεια τρίτης χώρας. Ε, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για πολύ σοβαρά δικαιώματα όπως είναι η διαφθορά, το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων όντων, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για το οργανωμένο έγκλημα και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό ο όρος διαφθορά να συμπεριληφθεί. Εγώ ξέρετε είμαι από την Πορτογαλία και αυτή τη στιγμή ο αντιπρόεδρος μιας πολύ κοντινή σε χώρας, της Αγγόλας, ε, πρέπει να απαντήσει στα πορτογαλικά δικαστήρια με κατηγορίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο για ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για απόπειρα παρακόλλησης της ε, διερεύνησης των κατηγοριών ξεπλύματος χρήματος και απόπειρα δωροδοκίας ε, των πορτογαλικών δικαστικών αρχών οι αρχές της Αγγόλας προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις διώξεις και επικαλούνται το γεγονό ότι ό,τι και να συνέβη, ακόμα και αν έχουν συμβεί αυτά, δεν έχουν συμβεί στην Πορτογαλία, έχουν συμβεί σε μια τρίτη χώρα. Όμως η διαφορά δικαστικού λειτουργού, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πάντοτε οδηγεί σε φυλάκιση γιατί ο συγκεκριμένο δικαστικός λειτουργός αποδείχθηκε και είναι στη φυλακή κτλ. Είναι λοιπόν απαραίτητο η νομοθεσία μας να είναι αποτελεσματική. Δεν ζούμε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Τα δίκτυα αυτά έχουν παγκόσμια δράση και πρέπει εμείς ε, να έχουμε διατυπώσεις πολύ σαφεί στη νομοθεσία μας. Και τέλος, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ένα τομέα στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, θα δούμε τις τροπολογίες που θα υποβληθούν, ένα τομέα που πιστεύω ότι επιδέχεται βελτιώσεων και πρέπει από εκεί σε αυτό να διδαχθούμε από τα ευρήματά μας για τα Panama Papers, είναι το εξής. Βασικοί παράγοντες αυτής της διαδικασίας ξεπλήματος χρήματος είναι επαγγέλματα τα οποία θα έπρεπε να υποχρεούνται από τον νόμο να αναφέρουν ότι έχουν υποψίες για τη διάπραξη αδικημάτων και αναφέρομαι δηλαδή σε δικηγόρους, σε λογιστές, σε εταιρείε κτηματομεσητικές. Κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί να ενισχυθούν οι ποινικέ κυρώσεις αλλά να μην περιοριστούμε στις ποινικέ κυρώσεις, αλλά να ενισχύσουμε τις διοικητικές κυρώσεις, αλλά και κυρώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή ή και ε, απόσυρση της άδειας ασκήσεως επαγγελματός. Συχνά αυτά τα επαγγέλματα υποτίθεται ότι ε, δίνουν λογαριασμό στην διοντολογία και στους φορείς διοντολογία των επαγγελματικών του συλλόγων και επαγγελματικών οργανώσεων. Όμως, στα Panama Papers και στη σχετική επιτροπή είδαμε ότι αυτό ε, δεν λειτουργεί τελικά. Το FIU και τα διάφορα FIU μας λένε ότι έχουν πολύ λίγες εκθέσεις από αυτά τα επαγγέλματα. Έχουν ένα σωρό εκθέσεις και αναφορές από τις τράπεζες, γιατί το χρήμα όλο και περισσότερο ακολουθεί μια ροή χρηματοπιστωτική και τραπεζική, αλλά η δικηγορική σύλλογη, ε, τα σώματα ορκωτών ελεγκτών και το καθεξής, οι ενώσεις που τους εκπροσωπούν, δεν λαμβάνουν καθόλου τέτοιου είδους αναφορές. Εκεί γίνεται ένα τεράστιο πάρτι και ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και να υπάρξουν κυρώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αναιρείται, θα αναστέλλεται ή θα ακυρώνεται η άδεια σκήσεως επαγγέλματος και άρα θα υποχρεωθούν να αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Δεν ξέρω αν ο Ιγνάτσιο θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Εάν όχι, να ζητήσω από την Επιτροπή ο κύριος Μπλούμσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη δυνατότητα να αντιδράσω στο θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας, τον κύριο Κοράο, για το θάρρο και τη δουλειά που έχει κάνει τώρα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη φάση των συζητήσεων δεν μπορεί να πάρει θέση πέρα των τροπολογιών ή κατά, αλλά η πρώτη αποτίμηση των εμπειρογνωμόνων μας είναι πολύ θετική και ανυπομονούμε να συζητήσουμε περαιτέρω τις τροπολογίες μαζί σας. Ε, ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για τη στήριξη του προ τα βασικά στοιχεία τη πρόταση τη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, το αυτοπλήσιμο, την αυτονομιμοποίηση, όταν κάποιο ο ίδιος ασχολείται με την νομιμοποίηση των εσόδων του, γιατί τι περισσότερες φορέ τα από το έγκλημα, το, από το οργανωμένο έγκλημα, δεν ορίζεται έτσι και θα πρέπει να τιμωρείται από όλα τα κράτη-μέλη. Επίση, θα πρέπει όλα τα σοβαρά αδικήματα και εγκλήματα να αντιμετωπίζονται παρόμοιω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στιγμή κάποιοι φραγμοί από την νομοθεσία των κατώμελων που δεν επιτρέπουν τη διακριτική συνεργασία ω τώρα και αυτοί πρέπει να έρθουν. Ελπίζουμε το Ευρωκοινοβούλιο να καταλήξει μια κοινή θέση σύντομα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που κατά πάσα πιθανότητα θα στηρίξει τη θέση αυτή τη πλειοψηφία σας. Αυτό θα επιτρέψει να περάσουμε σε συζητήσεις και να νομοθετήσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Κύριε Κοράο, τη δική σας άποψη. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς, και οι παρατηρήσεις της συναδέλφου Χολμάγερ και της κυρίας Γκόμες είναι προτάσεις από τον οποίο συμφωνώ και στα στοιχεία αυτά νομίζω ότι θα βρούμε οπωσδήποτε λύση συμβαστική. Οπωσδήποτε για τον κατάλογο λόγου χάρη. Όταν έκανα την, καταλο... την παρουσίαση προηγουμένω με τα παραδείγματα δικημάτων, εγκλήματων, μίλησα για τρομοκρατία, διαφθορά. Όμω στην τροπολογία 9 υπάρχει ένα κατάλογο αρκετά διεξοδικό και πολύ ευρύ. Οπότε εκεί έχουμε τη δυνατότητα να τον διευρύνουμε εφόσον θέλουμε. Να τον επεκτείνουμε μάλλον. Η ουσία είναι να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων. Ώστε να καλύψουμε το δυνατόν όλες τις μορφές. Τις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία νομιμοποίησης. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείε, στόχος είναι να ε, συμπεριλάβουμε και τα νομικά πρόσωπα. Είτε μικρών ή μεγαλύτερων διαστάσεων, δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς αυτό, ή αρμόδιες αρχές θα πρέπει. Και οι ανακριτές των διαφόρων κρατών, εκείνοι θα τα εντοπίσουν για τις παρατηρήσεις της συναδέλφου Γκόμες Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να ενισχυθεί τόσο η δικαστική συνεργασία όσο και κάθε είδους ε, βάσει της οδηγίας που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε και ένα σύστημα ποινών ώστε για το περιεχόμενο της οδηγίας ναι, έχει μια αποτελεσματικότητα κάποιες φορές. Αρκούν οι διοικητικές, ή αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές για να διακοπεί μια δραστηριότητα, αλλά όχι μόνο. Πάντως και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι στο ίδιο μήκος βρισκόμαστε. Θα προσπαθήσω την πρόταση να τη βελτιώσω, την πρόταση οδηγίας. Να γίνει στο το δυνατόν σαφέστερη και αποτελεσματική. Αυτό είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι με τις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών και με την επεξεργασία τροπολογιών θα πετύχουμε ακριβώς αυτό το στόχο όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την ε, πολύ σοβαρή δουλειά σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Να αναφέρω ότι η προθεσμία την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Οκτωβρίου στις 12. ώστε να έχουν αρκετό χρόνο όλες οι ομάδες. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 19 Οκτωβρίου και θα προλάβουμε να έχουμε και μεταφράσεις χάρη στην παράταση της προθεσμίας. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι στις 13 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Και πάμε αλλού, σε άλλο σημείο. 15, 16, 17. ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο για την 7η ε, έκθεση πρόοδου σε σχέση με την υλοποίηση της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επίσης, ε, συντονιστής τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση για την 14η έκθεση της μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απόφαση κοινή στις δύο υποθέσεις ε, για, από τις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και για τις προσφυγές της Σλοβακίας και Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού για την υποχρεωτική επανεγκατάσταση ετούντων άσυλων. Συνάδελφοι, Είναι οι δύο λοιπόν αυτές αποφάσεις κατά και απόφαση για την επανεγκατάσταση 160.000 ατόμων από την Ιταλία και την Ελλάδα και να βοηθηθούν αυτά τα κράτη-μέλη να χειριστούν τις μεγάλες ροές ανθρώπων που ζητούν διεθνή προστασία ζητούσαν μάλλον πριν δύο χρόνια τον το Συμβούλιο ενέκρινε τι διαφορέ αυτέ, ε, διεθνή προστασία. Τον Ιούλιο 2015 το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να επανεγκαταστήσει 22.504 ανθρώπου από χώρε που είχαν πάρα πολλού πρόσφυγε λόγω τη κρίση στη Συρία. Σήμερα, δύο μέρε πριν την εκπνοή των αποφάσεων για την επανεγκατάσταση, σημειώνουμε ότι 20.000 άτομα επανεγκαταστάθηκαν αποτελεσματικά από την Ελλάδα και λιγότεροι από 9.000 από την Ιταλία. Ενώ 17.000 θα έπρεπε να έχουν ε, μετακατασταθεί, ιδίω από την Τουρκία. Οι αριθμοί δείχνουν από τη μια ότι οι προσδοκίες του 2015 δεν έγιναν σεβαστές, δεν επετεύχθησαν, αλλά από την άλλη η μετεγκατάσταση και η επανεγκατάσταση μπορούν να λειτουργήσουν. Η δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που ενισχύει το επίπεδο συνεργασία με την Τουρκία και συμβάλλει στη μείωση αφήξεων στην Ελλάδα δεν αρκεί. Ένας άλλος λόγος για την έλλειψη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου είναι η άρνηση των κρατών μελών να συνεργαστούν. Δύο κράτη-μέλη έχουν προσφύγει κατά των αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως το Δικαστήριο απέρριψε τις αξιώσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας πριν από λίγες μέρες. Θα ακούσουμε μία ε, σύνοψη της απόφασης από την νομική υπηρεσία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έριξε δικασίες παραβάσεις παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Πολωνίας, διότι οι τελευταίες χώρες δεν έχουν μετακαταστήσει κανέναν ε, με αυτό το συνολικό, το, μέσα σε αυτό το συνολικό τοπίο θέλω να ακούσουμε την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με την επικατάσταση και κατάσταση καθώς υπάρχουν ακόμη άτομα επιλέξιμα για το σύστημα μετακατάστασης, ιδίως στην Ελλάδα, και ε, η ανάγκη για μετακατάσταση από τις χώρες της Νοτήρης Μεσογείου έχει μεγαλώσει. Κύριε Φερβέ, Έχετε το λόγο για να μας δώσετε την ενημέρωσή σας για τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Για τη δήλωση αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μπορώ να πω ότι συνεχίζει να αποφέρει αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους έτσι όπως αυτοί διατυπώθηκαν από τους επακεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την αύξηση των αφήξεων τους τελευταίους μήνες, οι αφήξεις παραμένουν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι πριν έχουμε τη δήλωση αυτή. Από τότε που άρχισε να ισχύει η δήλωση έχουμε κατά μέσο όρο 80 αφήξεις καθημερινά, ενώ έχουμε 4.000 την ημέρα αφήξεις 6 μήνες νωρίτερα. Πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή σας έχει συζητηθεί το θέμα των θανάτων των ανθρώπων αυτών. Θάνατοι έχουν μειωθεί κατά πολύ, αντίστοιχα με τη μείωση στον αριθμό των αφήξεων. Τώρα για να δούμε τα βασικά στοιχεία. Η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου έχει προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά. Μέχρι τώρα οι υπηρεσίε ασύλου που στηρίζονται από την ΙΑΖΟ έχουν επεξεργαστεί 25.000 τέτοιες αιτήσει σε πρώτο επίπεδο και σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα δράσης που συμφωνήσαμε με τον Υπουργό Μουζάλα, τον Ιούνιο φέτος η καθυστέρηση που υπήρχε σε αυτή την ε, πρώτη επεξεργασία, σε πρώτο επίπεδο, είχε καλυφθεί. Δυστυχώς και εξαιτία των αυξήσεων ε, στις ε, αφήξεις, δυστυχώς εμφανίστηκε και πάλι καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτήσεων αυτών και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Πάντως πιστεύω ότι με κοινή δράση από την ΕΖΟ, τις υπηρεσίες ασύλου, θα μειωθεί η καθυστέρηση αυτή και πάλι και θα καλυφθεί. Είναι πολύ σημαντικό οι χώρες μέλη να συνεχίσουν να στέλνουν τους εμπειρογνώμονές τους, τους ειδικού τους, μέσω της ΙΑΣΟ. Για να σας δείξω πώς λειτουργεί το πράγμα, 370 σήμερα εργάζονται στα νησιά για να χειριστούν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με αιτήσει ασύλου. Διερμηνείς, ειδικού και άλλους αξιωματούχους. Πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή σας επίσης αναφέρθηκε το αδιέξοδο όσον αφορά την απόφαση που λαμβάνεται σε δεύτερο επίπεδο εξέτασης των αιτήσεων. Δυστυχώς, εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Όπως έχω πει και άλλες φορές, 13 επιτροπές δημιουργήθηκαν όταν ήταν σαφές ότι η παραγωγικότητα της ε, μιας δεν ήταν ικανοποιητική, μπαίνανε άλλοι με μέσα πληροφορικής, με στήριξη. Παρόλα αυτά όμως η απόδοση δεν έχει βελτιωθεί. Και έχουμε ακόμα επεξεργασία 30 υποθέσεων τη βδομάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ λίγο. Πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, στο Συμβούλιο μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθε απόφαση για δύο Σύριους που είχε αποφασιστεί να επιστραφούν στην Τουρκία. Το State Council αποφάσισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να επιστραφούν. Οπότε ανεστάλλει η απόφαση. Βάση της περίπτωσης αυτής ίσως τελικά να βοηθηθούν οι αρμόδιοι που παίρνουν την απόφαση και να μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να παίρνουν τις σχετικές τους αποφάσεις βασιζόμενες σε αυτό το παράδειγμα. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με αυτό είναι οι επιστροφές που είναι λίγες αλλά γίνονται από την αρχή της δήλωσης 925 έχουν επιστραφεί στην Τουρκία. Πρόκειται κυρίως για επικόους τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. 200 Σύριοι επίσης έχουν επιστραφεί αλλά σε θελοντική βάση. Αποφάσισαν δηλαδή να επιστρέψουν. Το άλλο τώρα που γίνεται κατάφορο είναι ότι η ελληνική αστυνομία αντιμετωπίζει προβλήματα προκειμένου να εντοπίσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει αποδέκτες μιας αρνητικής απόφασης για την περίπτωσή τους. Και πράγματι όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται να καταλήξουν ευχές σε απόφαση, ε, τόσο πιο δύσκολο είναι μετά να βρεθούν και άνθρωποι που τους αφορούν οι αποφάσεις αυτές. Πρέπει η διαδικασία να είναι δίκαια βέβαια, αλλά πρέπει να είναι και ταχεία. Δηλαδή να μην πρέπει ο κόσμος να περιμένει υπερβολικά πολύ μέχρι να έχει μια απάντηση. Συγχρόνω, βέβαια πρέπει να καταλάβει κανείς τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όσο περιμένουν, πού βρίσκονται, πού κυκλοφορούν, να έχουμε πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια διαχείριση δεδομένων. Και τέλος, ξέρω ότι δεν είναι κάτι πολύ δημοφιλέ εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά έχει να κάνει με την αποτελεσματική πολιτική επιστροφών πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι θα επιστρέψουν που αποφασίζεται είτε πρόκειται για τη Λέσβο, είτε πρόκειται για αλλού, η δυνατότητα αυτή βοήθειας προς αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μεγάλη, δυστυχώς. Όσον αφορά τώρα τις εθελοντικές επιστροφές, αυτές λειτουργούν ικανοποιητικά. Σας είπα, 200 Σύριοι επέστρεψαν βάσει αυτού και 800 απευθείας από τα νησιά. Και φτάνω στο πιο δύσκολο σημείο, που είναι ότι εξαιτία της αύξησης των αφήξεων που διαπιστώσαμε τους τελευταίους δύο μήνες, οι συνθήκες τους καταβλισμούς, παρόλο που είχε πάρεξει κάποια βελτίωση πριν, Τώρα ξανά βρισκόμαστε στην κατάσταση όπου είναι υπερβολικά πολυάριθμοι όσοι βρίσκονται στους καταβλισμούς στη Λέσβο και στη Σάμο κυρίως. Μεγάλη συγκέντρωση. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Για να μην υπάρχει όμως παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι όλοι κρατούνται. Το ακούτε αυτό καμιά φορά. Αν δείτε όμως τα νούμερα, πόσοι φτάνουν Από την άλλη, οι γεωγραφικοί περιορισμοί έχουν αρθεί. Πάντως η πίεση στα νησιά αυξάνει πάλι. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλη πρόκληση. Θα προσθέσω κάτι αργότερα, ίσως με τα σχόλια. Πάντως το τελευταίο που θέλουν να πω τώρα και είναι μια πιο θετική χρειά όσον αφορά την υπηρετική χώρα. Εκεί η κατάσταση βελτιώνεται από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που είχαμε στην αρχή, όταν άρχισε να υλοποιεί τη δήλωση, τώρα μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχουν οι διευκολύνσεις, υποδομές, επειδή το πρόγραμμα μετακατάστασης προχωράει κάπως πιο γρήγορα εξαιτίας ε, της μετακίνησης σε θελοντική βάση κτλ δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καθόλου προβλήματα. Στην επιρωτική χώρα επίσης εποφελούνται οι άνθρωποι και από κάποια ποσά σε ρευστό που παίρνουν, κάτι το οποίο τους βοηθά να διαθέτουν κάποια αυτονομία. Οπότε η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στην υπηρετική χώρα από ό,τι στα νησιά. Για την ε, μετεγκατάσταση θα σας τα πει βέβαια ο κύριος Νίλσεν, αλλά εγώ ένα πράγμα θέλω να αναφέρω εδώ για την Ελλάδα. 66.000 θα έπρεπε να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και μόνο 20.000 έχουν μετεγκατασταθεί. Εδώ θέλω να τονίσω και το έχω πει και παλιότερα ότι αυτές 66.000 είναι ένα νούμερο που αποφασίστηκε πριν αρχίσει να ισχύει δήλωση με την Τουρκία. Δεν ε, υπήρχαν αυτοί 66.000. Οπότε προσοχή λίγο για τα συμπεράσματα στο οποία καταλήγει κανείς. Θα σταματήσω εδώ και σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις και θα έχω την ευκαιρία να επανέλθω αργότερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριο Νίλσεν, έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε για την μετεκατάσταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Ήδη αναφέρατε, Πρόεδρε, τους βασικούς αριθμούς. Θα φτάσουμε σε ένα σύνολο 30.000 που θα μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και την Ιταλία συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε περίπου 2.000 μετακαταστάσεις ε, το, το μήνα, ε, σε Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια μικρή πτώση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά σχετικά καλά. 6 Σεπτεμβρίου, 15η έκθεση, ήδη μιλούσαμε για το συνολικό αριθμό, βελτιώσαμε τις διαδικασίες, το σχεδιασμό γενικώ και σας επισημάναμε το τι συμβαίνει γενικώ με την μετακατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε κάθε περίπτωση τώρα σε σχέση με το τι θα γίνει στο μέλλον, κατά πρώτον πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου αυτές συνεχίζουν να ισχύουν για όσους φτάσουν ως την ελληνική επικράτεια στις 26 Σεπτεμβρίου. Όσους έφτασαν λοιπόν. Η πρώτη προτεραιότητα για μας είναι ότι όλοι οι αναπομείναντες μέχρι την ημερομηνία εκείνη που πληρώνουν τις προποθέσει και είναι επιλέξιμοι για την ε, μετεγκατάσταση και τους προτείνει η Ελλάδα και η Ιταλία θα μετεγκατασταθούν τους επόμενου μήνες εφόσον συνεχίσουν να υπάρχουν αιτήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τους ερχόμενους μήνες δηλαδή. Η εκτίμησή μα βάσει τη τωρινή κατάσταση και του αριθμού των ανθρώπων που έχουν καταγραφεί για με είναι ότι θα έχουμε περίπου 6-7 επιπλέον άτομα που θα πρέπει να μετακατασταθούν από την Ελλάδα συνολικά τους ερχόμενους μήνες, οπότε εκεί και θα εκπνεύσουν τελείως τα προγράμματα μετακατάστασης. Πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προτείνει παράταση της απόφασης διότι θέλουμε να αποστείλουμε το ισχυρό μήνυμα ότι τώρα οι συνομοθέτες πρέπει να προοδεύσουν στο Δουβλίνο για να περάσουμε από τα προσωρινά και επιτόπια συστήματα στην πραγματική αντιμετώπιση της κρίσης. Να υπάρχει κάτι δομικό, διαθετικό ως λύση. Και εκεί να προβλέψουμε υποχρεωτικούς και δεσμευτικού κανόνε για την κατάσταση ε, ώστε να είναι ε, ισχυρό το σύστημά μα στο μέλλον χωρί να βασίζεται σε προσωρινέ λύσει. Πέραν του συστήματο. Όπω είπαμε με την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε, δηλώνεται ότι. Μάλλον απευθύνεται έκκληση προ τα κατημέλη να συνεχίσουν επί την αλληλεγγύη προ την Ιταλία και την Ελλάδα μέχρι να, να, μέχρι να αρχίσει να ισχύουν ο κανονισμό του δουπλίνου. Και να εκφράσουν και δύο αυτέ χώρε τη ίδια αλληλεγγύη χρειάζονται τι υπόλοιπε χώρε. Η έκθεση τη 6η Σεπτεμβρίου δεν απαιτεί έκθεση, βολιδο, έκθεση αποτίμησης ή ενημέρωσης για τα μαθήματα και τα διδάγματα που αντλήσαμε από όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι γνωστά από όλου. Το ανέφεραν όλε οι Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Το σύστημα αντικατάσταση μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να είναι αποτελεσματικό, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ώστε να ε, δείξει κανεί έμπρακτα την ε, αλληλεγγύη του προ τα κατημέλη αλλά για τα διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε, τις πρακτικές εμπειρίες όταν θέλουμε να προχωρήσουμε στο νέο σύστημα του Δουβλίνου, είναι πολύτιμα όλα αυτά. Για την επανακατάσταση είμαστε στις 23.000 άτομα, μετρώντας και τον Ιούλιο του 2015 με το σχετικό σύστημα και το τμήμα κατάσταση της Συμφωνίας Ελλάδας, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον Τουρκίας. Ως προς τα συμπεράσματα του 2015, τα συμπεράσματα του Ιουλίου του 2015, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ε, πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Για τα δύο προγράμματα, η χρηματοδότηση που προβλέπουμε για τα κράτη-μέλη αρχίζει να φτάνει στο τέλος της. Θα έχει εξελιχθεί στο τέλος της χρονιάς. Όπως ξέρετε, Έχουμε πρόταση για νέο πλαίσιο επανεγκατάσταση. Το εξετάζουμε, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Για να υπάρξει μετάβαση από το νέο σύστημα και το μελλοντικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε ε, δημοσιοποίησε μια σύσταση προ τα κατημέλη για 50.000 άτομα τα ερχόμενα δύο χρόνια. Αυτό συνοδεύεται με το ίδιο επίπεδο οικονομική στήριξη που ισχύει και τώρα, 10.000 ευρώ ανά άτομο που τον εγκαθίσταται. 500 εκατομμύρια ευρώ για την ε, επανακατάσταση για το διάστημα αυτό λοιπόν. 50.000 είναι ε, αριθμός ε, που έχουμε στόχο εμείς. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητε προποθέσει τουλάχιστον. Ελπίζουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό ή και ακόμη και καλύτερο. Και ακόμη καλύτερο αν τα κράτη-μέλη μα βοηθήσουν να πάμε παραπέρα. Υπάρχει και η σύσταση από την πλευρά μας, όπου θεωρούμε ότι η Ένωση πρέπει να ε, στοχεύσει τι προσπάθειές της, δηλαδή ε, οι χώρες από τις οποίες πρέπει να πάρουμε αυτούς 50.000 είναι η Τουρκία, η Ορδανία, η Λίβανο και 5-6 χώρες στην Αφρική που είναι είτε από τις μεγαλύτερες χώρες υποδοχή προσφύγων, είτε μέρος του δρόμου και των οδών που οδηγούν και καταλήγουν στη Λιβύη. Είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω σε ερωτήσει των συναδέλφων. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος, ε, η, κυρία Μωρίν από την νομική υπηρεσία. Παρακαλούμε να μας δώσετε στοιχεία για την περίπτωση της ε, Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εσείς το θυμήσατε. Η Σλοβακική Δημοκρατία και η Ουγγρική Δημοκρατία με δύο ξεχωριστά αιτήματα ζήτησαν την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου της 22 Σεπτεμβρίου 2015 που εγκαθιδρεί προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε με βάση το άρθρο 168 εδάφιο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου η Πολωνία παρενέβη υπέρ της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας ενώ Βέλγιο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Επιτροπή και άλλες χώρες ε, επενέβησαν υπέρ του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν παρενέβη σε αυτή την υπόθεση. Δεν παριστάθηκε. Το δικαστήριο απόρριψε τα δύο αυτά αιτήματα, τις δύο προσφυγές και είχε την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, να αποφανθεί για το σύνολο των μέσων που ε, υιοθέτησαν τα ε, κράτη που προσέφυγαν και άδραξε την ευκαιρία για να διευκρινίσει ενδιαφέροντα στοιχεία ε, και για τις διαθεσμικές σχέσεις αλλά και για τις διαδικασίες και τις αρχές που ε, υπάρχουν πίσω από την πολιτική σε θέματα ασύλου. Τα μέσα στα οποία προσέφηγαν τα κράτη που προσέφυγαν ήταν τριών ειδών. Πρώτον, το άρθρο 168 εδάφιο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρμόζει για νομική βάση της απόφασης ε, εναντίον της οποίας προσέφηγαν. Ένα άλλο, μια άλλη σειρά νομικών μέσων είχαν να κάνει με το κατά πόσο η διαδικασία λήψης της απόφασης ήταν σε εντάξει. Και μια, μια τρίτη σειρά νομικών μέσων ήταν επί της ουσίας, δηλαδή την αναλογικότητα του μέτρου αμφισβήτησαν. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην πρώτη σειρά νομικών επιχειρημάτων που έχει να κάνει με τη νομική βάση. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία σε γενικές γραμμές και κατά πρώτο λόγο στηρίζαν το εξή. Η νομοθετική και νομοπαρασκευαστική διαδικασία πρέπει να ισχύσει γιατί το άρθρο 168 εδάφιο 3 προβλέπει διαβούλευση με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προς αυτό, το δικαστήριο άδραξε την ευκαιρία για να υπενθυμίσει ότι μία νομική πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ω νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο εάν υιοθετείται με βάση συγκεκριμένη ρητή διάταξη της συνθήκης και αναφέρεται ρητός είτε σε ειδική νομοθεπαρασκευαστική διαδικασία είτε στη συνήθη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Στο άρθρο 168 δεν υπάρχει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθετική διαδικασία. Επομένως η απόφαση εναντίον της οποίας προσφεύγουν αυτά τα κράτη δεν αποτελεί νομοθετική πράξη που να πρέπει να υιοθετηθεί με την επίσημη οδό κατά τα λοιπά το δικαστήριο θεώρησε ότι το άρθρο 168 εδάφιο 3 επιτρέπει πράγματι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εθετήσουν όλα τα προσωρινά μέτρα που είναι απαραίτητα για να απαντήσουν με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο σε μια κατάσταση κατεπήγοντος η οποία διαμορφώνεται με την μαζική ξαφνική εισρωή εκτοπισμένων ατόμων και υπ' αυτή την έννοια τα προσωρινά μέτρα μπορούν να δώσουν λαβή για παρέκκληση παρέκκληση από την νομοθετική πράξη. Δηλαδή, ε, για να υπάρχει αυτή η παρέκκληση να μην υιοθετηθεί η νομοθεσία αλλά προσωρινή, ε, προσωρινό μέτρο, θα πρέπει να ε, περιορίζεται στο χρόνο και στο χώρο ως προς το πεδίο εφαρμογής. Και να μην έρχονται αυτά τα προσωρινά μέτρα να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν μονίμως τις, νομ, τα, τις νομοθεσίες από τις οποίες προβλέπουν παρέκκληση και θεωρεί το δικαστήριο ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής το προσωρινό χρονικά, δηλαδή από 22 Ενάτου 15 μέχρι 26 Ενάτου 2017. Αυτό ε, σύμφωνα με το δικαστήριο ορίζεται σαφέστατα, άρα ο προσωρινός χαρακτήρας του μέτρου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όταν ρητός αναφέρεται η προθεσμία, το χρονικό διάστημα στο οποίο ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο. Στη συνέχεια η Σλοβακία θεώρησε ότι μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι οι προϋποθέσεις, δηλαδή το κατεπήγον σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, ε, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυτές για να προσφύγει κανείς τα προσερινά μέτρα. Ερχόμαστε τώρα στο τυπικό. Προσέφηγαν και εναντίον του τυπικού της διαδικασίας. Οι δύο χώρες που προσέφυγαν επικαλέστηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 25-26 Ιουνίου που είχαν προβλέψει ε, τη διαδικασία της επίγουσας μετεγκατάστασης και το Συνδικαστήριο σημειώνει ότι κατά τα λοιπά αυτά είχαν ήδη γίνει με μια πρώτη απόφαση μετεγκατάστασης που είχε υιοθετήσει το Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου του 2015 που αναφερόταν σε 40.000 ανθρώπους που ζητούσαν διεθνή προστασία και ε, βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Επομένως, οι δύο προσφεύγουσες χώρες υποστήριζαν ότι ε, η απόφαση ξεπερνάει το πεδίο εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και άρα δεν τηρούσε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου γιατί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είχαν προβλέψει ότι η απόφαση εγκατάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται με συνένεση. Και ε, η απόφαση είχε ληφθεί με ειδική πλειοψηφία. Υπ' αυτή την έννοια το δικαστήριο πρώτα επεσήμανε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είχαν ήδη εφαρμοστεί μέσα από άλλη απόφαση την προηγούμενη του Σεπτεμβρίου 2015 και όχι ε, μέσα από την απόφαση εναντίον της οποίας προσέφυγαν οι δύο χώρες και σύν της άλλης οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να στερήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα ίδιας πρωτοβουλίας που έχει. Επομένως, ακόμα και αν δεν είχε προβλεφθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης για άλλους ανθρώπους και πέραν από τους 40.000 ανθρώπους για τους οποίους υπήρχε η πρώτη απόφαση, τίποτα δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με την κατάσταση για άλλους ανθρώπους, το οποίο και έπραξε άλλωστε. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξουν οι κανόνες ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 73 και προβλέπουν την ειδική πλειοψηφία. Κατά τα λοιπά, οι δύο αυτές χώρες αναφέρθηκαν στο ότι καταστρατηγήθηκε η υποχρέωση το Συμβούλιο να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι αυτό πρέπει να υπερισχύσει. Και ε, θεωρήθηκε ότι μπορεί να υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις έναντι της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι το οποίο ωφελούσε βασικά την Ελλάδα, την Ιταλία αλλά και την Ουγγαρία. Εν τω μεταξύ η Ουγγαρία έχει ζητήσει να εξαιρεθεί, να αποσυρθεί, να μην ωφεληθεί πλέον από τη συγκεκριμένη απόφαση και άρα η νέα απόφαση δεν αφορούσε πλέον την Ουγγαρία και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο. Σύμφωνα λοιπόν από την Ουγγαρία και την Σλοβακία, ε, όταν δεν ξαναγίνεται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, επειδή αποσύρθηκε η Ουγγαρία, αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο παρέλειψε να διαβουλευτεί το Κοινοβούλιο και άρα ε, παραβαίνει και καταστρατηγεί την υποχρέωση. Επειδή στη δεύτερη απόφαση εξαιρέθηκε ένα από τα μέλη και αποσύρθηκε. Θεώρησε λοιπόν το ε, δικαστήριο ότι η μη τήρηση αυτών μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση ε, του, της νομοθετικής πράξης. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοιχεί στην αποτελεσματική συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, θεσμικής ισορροπίας στην οποία αποσκοπούν οι συνθήκες και αποτελεί έκφραση της δημοκρατικής ελευθερίας των λαών, τη συμμετοχή στην εξουσία. Το δικαστήριο λοιπόν υπενθυμίζει αυτή την αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι η απόφαση που υιοθετήθηκε τελικά από το Συμβούλιο απόκλινε στην ουσία της από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι δεν λαμβανόταν πλέον ε, προς όφελος και της Ουγγαρίας. Ωστόσο, και τούτων λεχθέντων, το δικαστήριο αυτό το παραδέχεται, ωστόσο διαπιστώνει ότι το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε δεόντως για αυτή την τροποποίηση από την Προεδρία του Συμβουλίου στην έκτακτη συνεδρίαση του Ισολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Σεπτεμβρίου του 2015 πριν εγκρίνει το ψήφισμά του. Άρα το Κοινοβούλιο είχε την ευκαιρία στο ψήφισμά του να είχε λάβει υπόψη του τις τροποποιήσεις που του ανακοινώθηκαν από το Συμβούλιο. Άρα ήταν δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο και το δικαστήριο ολοκλήρωσε το σκεπτικό του λέγοντας ότι τα λοιπά μέτρα δεν αλλίωσαν την ουσία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα δεν απαιτεί το εκ νέου διαβούλευση με το Κοινοβούλιο λόγω αυτού. Τώρα, οι δύο αυτές χώρες ε, Επίσης προέβαλαν τα εξής επιχειρήματα, τους νομικούς ισχυρισμούς. Το Συμβούλιο είχε τροποποιήσει επί της ουσίας την πρόταση της Επιτροπής χωρίς να αποφασίζει ομοφόνος βάσει του άρθρου 293 δάφιο 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε de facto τροποποιήσει την αρχική της πρόταση από τη στιγμή που εγκρίνει τις τροποποιήσεις του κειμένου αυτού με τις διάφορες συνεδριάσεις ε, των ομάδων του Συμβουλίου και άρα δεν υπήρχε πλέον ανάγκη να γίνει σεβαστή η αρχή της ομοφωνίας. Και τέλος, η απόφαση δεν αποτελεί νομοθετική πράξη και άρα η διαδικασία υιοθέτησης της απόφασης δεν υπόκειται στις απαιτήσει που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, αντιθέτως με ό,τι φρονούσαν οι δύο αυτές ε, χώρες. Και για να ολοκληρώσω, για τα θέματα για την τρίτη σειρά νομικών επιχειρημάτων που είχαν να κάνουν με την ουσία και κυρίως για την αναλογικότητα αυτής της απόφασης. Το δικαστήριο θεώρησε ότι ο μηχανισμός κατάσταση που προβλέπει η απόφαση εναντίον της οποίας προσέφηγαν οι δύο χώρες δεν συνιστά μέτρο που προδήλως δεν ταιριάζει στην επίτευξη του στόχου. Ε, στόχος ήταν δηλαδή να βοηθηθεί η Ελλάδα και η Ιταλία να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση του 2015. Άρα αναδρομικά. Δεν μπορεί κανείς αναδρομικά να έρχεται να λέει ότι ένα μέτρο ήταν δυσανάλογο προς την αποτελεσματικότητά του. Ο νομοθέτης, όταν νομοθετεί, προβαίνει για συγκεκριμένες εκτιμήσεις και αυτές οι εκτιμήσεις αμφισβητούνται ε, εκ των υστέρων μόνο όταν ήταν γνωστό ότι πάνω σε εσφαλμένα συμπεράσματα βάσισε τις εκτιμήσεις του και τις αποφάσεις του τη στιγμή που τις υιοθέτησε. Δηλαδή, το Συμβούλιο έκανε λεπτομερή εξέταση των στατιστικών στοιχείων που ήταν διαθέσιμα τότε, ανάλυσε αντικειμενικά τις επιπτώσεις με τα υφιστάμενα ε, στοιχεία τότε και τα οποία δεν ήταν εσφαλμένα τότε, άρα εάν ε, εκ των υστέρων ε, διαπιστώθηκε ότι ήταν δυσανάλογη προσέγγιση, σε αυτό δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν υπάρχει δηλαδή έλλειψη αναλογικότητας το δικαστήριο σημειώνει το μικρό αριθμό των μετεγκαταστάσεων που έγιναν μετά από αυτή την απόφαση και αυτό εξηγείται από μια σειρά στοιχείων τα οποία το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τη στιγμή που υιοθέτησε αυτή την απόφαση και οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας κυρίως από κάποια κράτη-μέλη. Επομένως, αφορτιόρι, ε, το Συμβούλιο δεν μπορούσε να περιμένει ότι δεν θα υιοθετούνταν ε, ε, αυτά στη συνέχεια. Όταν ε, σε κάθε περίπτωση ε, τα ε, οι στόχοι αυτοί δεν θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί με, λιγότερα, με λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Ο μηχανισμός που προβλέπεται από την πρώτη απόφαση μετεγκατάστασης είναι κάτι που δεν θα αρκέσει αυτό για να αντιμετωπίσει κανείς τη ροή, το, τη μεταναστευτική τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015. Σύμφωνα με το δικαστήριο, το Συμβούλιο θεώρησε ότι ο δεσμευτικός ε, χαρακτήρας επιβάλλεται λόγω του επίγοντος της κατάστασης. Είναι σημαντικό να σημειώσει κανείς ότι το δικαστήριο συνδέει αυτό το θέμα με την αρχή της αλληλεγγύης, άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό επιβάλλεται βάσει του άρθρου 80 και ήταν υποχρεωμένο να το λάβει αυτό υπόψη. Δικαστήριο επίσης όσον αφορά την Ουγγαρία και τη δικιά της την περίπτωση εκτίμησε έκανε, πρέβησε μία ανάλυση των διαφόρων μηχανισμών διόρθωσης που προβλέπονται από την πράξη και βάσει των μηχανισμών αυτών μπορούσε αναλογικά να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση σε κάθε χώρα μέλος. Στο ίδιο πνεύμα στην περίπτωση της Πολωνίας, στην ε, παρέμβασή της η Πολωνία είπε ότι οι χώρες μέλη περίπου ομοιογενώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν παραπάνω βάρος για να δεχτούν τους μεταγκαστημένους. Το δικαστήριο λοιπόν είπε ότι το επιχείρημα αυτό είναι απαράδεκτο γιατί ξεπερνάει αυτό το οποίο παρουσίασε ο βασικός παράγοντας η Ουγγαρία και έτσι λοιπόν για την περίπτωση της Πολωνίας είπε ότι μία μετεγκατάσταση η οποία θα εξαρτηθεί από πολιτιστικούς ή γλωσσικούς δεσμούς του ετούντος διεθνή προστασία και την χώρα προς μετεγκατάσταση οδηγούσε σε δυναμία τελικά κατανομής των ανθρώπων αυτών βάσει της αρχής της αλληλεγγύης και το δικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον ληφθεί υπόψη αυτός ο ε, παράγοντας καταγωγής αντιβαίνει στην ε, Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απέρριψε το δικαστήριο τα περί σαφήνειας ή αβεβαιότητας και μίλησε για μη τήρηση της αρχής της Γενέβης. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για τις πλήρεις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν βλέπω τους κύριους Σκέλλερ και ε, Πιόρ που είναι εισηγητές. Συζήτηση λοιπόν. Και ίσως οι συντονιστές. Όχι. Α, η Σόφιν Χετφέλτ. Εσείς ζητήσατε πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν περίμενα να μου δώσετε το λόγο τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Έχω πολλές ερωτήσεις. Κυρίως όσον αφορά τους δύο πρώτους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που ακούω ότι η Επιτροπή επιμένει πολύ επί των δύο νομοθετών και κυρίως επί του Συμβουλίου να πιέσει και αυτό για την τροποποίηση του συστήματος του Δουβλίνου. Αυτό επίγει. Αλλιώς θα προχωράμε από τη μία κατεπίγουσα λύση στην άλλη. Τώρα κατά τα άλλα για τη δήλωση με την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο δεν είπατε είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και η κατάστασή τους. Ένα μέρος της δήλωσης ήταν ότι δίνουμε πολλά χρήματα στις τουρκικές αρχές για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Πώς ελέγχεται την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε ότι έχουν φτάσει διάφορες εκθέσεις για βία, για παιδική εργασία, για διασμούς, ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και αναγκάζονται να επιστρέψουν στη Συρία πολύ. Εσείς πώς ελέγχετε το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε βεβαθεί ότι όλα τα παιδιά, ας πούμε, πάνε σχολείο στην Τουρκία τώρα. Και αν... Ναι, πώς. Και αν κατάλαβα καλά, είπατε 1925 επιστροφές υπήρξαν στην Τουρκία. Αν όμως δω τι μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί στην Τουρκία, έχετε υπολογίσει πόσο κοστίζει κατά κεφαλή η επιστροφή αυτή. Είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός για να τα περνάμε τα χρήματά μας. Και έπειτα ακούμε ότι χρησιμοποιούν εναλλακτικέ διόδους οι άνθρωποι για να πάνε ας πούμε στη Ρουμανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα και γι' αυτό. Είπατε ότι πολλοί είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά. Εμείς ακούμε ότι αυξάνονται οι εντάσεις, ότι οι συνθήκες του συνάθλιες ακούμε για όλο και περισσότερους που υποφέρουν από στρες, άγχος. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα και γι' αυτό. Και τέλος, πέρα από την υλοποίηση της δήλωσης με την Τουρκία. Μήπως ανησυχείτε εσείς ποτέ για το τι θα γίνει αν ετούντε άσυλο και πρόσφυγε μαζικά ε, φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να μην είναι πια τόσο χαρούμενη και επί ή που θα πρέπει να επιστρέψουν ή αλλιώς εμείς δεν σας λύνουμε το πρόβλημά σας. Ευχαριστούμε. Με κύριε Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή δεν ήθελα να πάρω το λόγο γιατί ναι με ειλικρινής ακούμε τα ίδια και πάλι ακούσαμε τα ίδια και τα ίδια. Και ένα από τα πράγματα που εμείς λέμε και ξαναλέμε είναι ότι χώρες μέλη οι υπερβολικά πολλές χώρες μέλη δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν δίνουν τα χρήματα ούτε για το αφρικανικό καταπίστευμα για να βοηθεί η κατάσταση αυτή την Ήπειρο, ούτε τεχνικό εξοπλισμό για να βελτιωθεί το έργο της ΙΑΖΟ και της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Έχω βαρεθεί πια. Εν πάση Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις για την κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά τους πρόσφυγες. Έχετε σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των προσφύγων που ήταν στην Τουρκία πριν αρχίσει να υλοποιείται η δήλωση και ξέρουμε πόσοι είναι οι πρόσφυγες στην Τουρκία σήμερα. Έπειτα δίνουμε πολλά χρήματα στην Τουρκία για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Πάντα όμως γνωρίζαμε ότι λίγοι είναι οι πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στους καταβλισμούς. Οπότε ποιος παίρνει τα χρήματα αυτά και για τι σκοπό και πόσοι είναι οι πρόσφυγες που βρίσκονται σε καταβλισμούς σήμερα. Και έχουμε καθόλου πληροφορίες για το αν ομάδες προσφύγων τυχαίνουν διαφορετικής μεταχείρισης στην Τουρκία ή μπορούν όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να πάνε σχολείο, τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Και τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. Για το θέμα της απόφασης για, τη μετακόμη, για την ε, μεταγκατάσταση. Ε, χαίρομαι που λέει η Επιτροπή θα συνεχίσει με τα νούμερα που έχουμε αποφασίσει, αλλά μπορείτε να μας πείτε αν συνεχίσουμε με τα νούμερα που έχουμε μέχρι τώρα στον αφορά την μετεγκατάσταση πόσοι μήνες ή χρόνια θα χρειαστούν ώστε 160.000 να έχουν μετεγκατασταθεί. Ευχαριστώ επίσης και τον συνάδελφο που εξήγησε την απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την προσφυγή της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας. Βεβαίως και όλοι γνωρίζουμε το αποτέλεσμα ε, της απόφασης που ήταν εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως ήταν καλό να τα ακούσουμε. Εγώ δεν ήξερα το εξή. Πόσο ανήσυχος είναι ένας από αυτούς, ο Ορμπάν, για παράδειγμα, που ανησυχεί που τα δημοκρατικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου του δεν τηρούνται. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και το ερώτημα είναι, οι χώρες αυτές τώρα θα τηρήσουν, θα σεβαστούν την απόφαση και όχι μόνο στα χαρτιά, θα πάρουν πρόσφυγες τέλος πάντων. Και έχουμε κάποια πληροφορία από τις γύρω χώρες μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βερζιάτα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με την κόποση που ξέφρασε ότι έχουμε η σας. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε οι κυρώσεις να είχαν επιβληθεί στις χώρες αυτές και πολύ νωρίτερα. Ε, η Κομισιόν όμως δεν το κάνει ξεκινάει μια διαδικασία επί παραβάση απέναντι σε τρεις, αλλά δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να έχει τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στη μετεγκατάσταση. Και αν κατάλαβα καλά τα νούμερα, πέρα από το θέμα της Τουρκίας, είμαστε σε λιγότερο από 30.000 μετεγκατάσταση από Ιταλία και Ελλάδα. Αυτή που είναι από την Τουρκία δεν είναι μετακατάσταση, είναι επανεκατάσταση εφόσον δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεδομένη τη κατάσταση Τουρκία, στην Τουρκία δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Μια στιγμή να συγκεντρωθώ. Α, ναι, λοιπόν, αν μετράω καλά, το 1 τέταρτο των υποχρεώσεών του έχουν φέρει σε πέραση χωρί μέλη. Και η Κομισιόν, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, θέλει να αποφύγει τη διόνυση αυτής της κατάστασης και περιμένει την υποτιθέμενη συμφωνία, θα έλεγα, υποτιθέμενη, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα αλλάξει κάτι. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι 6-7 άνθρωποι ακόμα θα υποφεληθούν από τη μετακατάσταση και ότι θεωρείτε πως όποιος φτάνει στην Ιταλία στην Ελλάδα πριν από τις 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να υποφεληθεί από την μετακατάσταση. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Οι χώρες μέλη λένε ότι θέλουν να μετακατάσταση εγκαταστήσουν μόνο όσους φτάσανε πριν τη δήλωση με την Τουρκία. Αυτοί δικαιούνται τη μετεγκατάσταση. 6-7 χιλιάδες. Αν όντω 27 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία, ποιος τελικά μπορεί να αποφεληθεί από την μετεγκατάσταση. Και πάλι, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η ελληνική αστυνομία δυσκολεύεται να εντοπίσει αυτούς που θα έπρεπε να επιστραφούν στην Τουρκία. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Και ποιες είναι οι εθνικότητες των, ε, των ε, ανθρώπων οι οποίοι, λέτε, σε θελοντική βάση επέστρεψαν και σε σχέση με τους 1925 που επιστράφησαν προς την Τουρκία, ποια είναι η προέλευσή τους και πού έχουν καταλήξει. Κάτι που ρώτησε και άλλος πριν από μένα. Για τα χρήματα. Στην Τουρκία φαίνεται ότι βάζουν τα παιδιά σε καταναγκαστική εργασία. Τι ισχύει. Είναι αλήθεια. Και πώς το ελέγχεται. Επίσης η νέα μετακίνηση προς τα ελληνικά νησιά που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ξέρουμε για την Ιταλία, που εκεί μειώνονται οι αφήξεις. Και να σας ξαναπώ αυτό που έχω ξαναπεί την προηγούμενη φορά. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κινησμός εδώ και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη να λέμε ότι μειώνονται οι θάνατοι και να το συγκρίνεται αυτό με τον αριθμό των αφήξεων. Μη μας λέτε τέτοια. Είναι απαράδεκτο. Κυρίως όταν ξέρουμε ότι συνεχίζονται να αυξάνονται αυτοί οι θάνατοι στη Μεσόγειο δυστυχώς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Γιουρέκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του δικαστηρίου έχει ως έχει. Είναι ένα γεγονός και μπορεί κανείς να συζητήσει πολύ για την νομική βάση στην οποία βασίστηκε. Πάντως, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αξιολογούμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όσον αφορά το μεταναστευτικό κύμα που έλαβε χώρα μετά τον πόλεμο στη Συρία, εδώ δεν πρόκειται για φυσικές καταστροφές που δεν έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη δράση τότε όντω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αλληλεγγύη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πολιτική των χωρών μελών. Και αυτή η πολιτική η οποία οδήγησε σε αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Το ακούσαμε και στην ομιλία του κύριου Γιούγκερ, ο οποίος είπε ότι η μόνη λύση για να δοθεί διέξοδος στο μεταναστευτικό πρόβλημα είναι να ανοίξουν οι πόρτες στην νόμιμη μετανάστευση. Και στην συζήτηση που έγινε μετά, η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα στην οποία νίκη ουσιαστικά και ο κύριος Γιούγκερ, μας είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση. Λοιπόν, εδώ πρέπει να θυμόμαστε ποιο είναι το καθήκον μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι να αξιολογούμε την πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι με την απόφαση αυτή λύνεται το πρόβλημα. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βερζιά, η οποία άρχισε από μια αρχή, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από τη δικιά μου, αλλά είπε επίσης ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υλοποιούνται. 85% των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Αν λοιπόν δεν εφαρμόζονται, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, σημαίνει ότι είναι και στραβές. Αυτό πρέπει εμείς να αξιολογούμε. Και όχι η πλειοψηφία να προσπαθεί να επιβάλλει την αποψή της ή με νομικές αποφάσεις κτλ κάποια πράγματα δεν γίνεται να εφαρμοστούν. Η ε, κυρία Σίπερ. Ήθελα πολύ σύντομα μια παρατήρηση επιπλέον, μάλλον μια διόρθωση να κάνω. Εδώ, αν θέλαμε να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές παρά της ε, μετανάστευσης, χωρίς καμία εναλλακτική, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι δεν θα δεχόμαστε κανέναν απολύτως πρόσφυγα. Δηλαδή δεν θα εκπληρούσαμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις να προσπαθήσουμε να ε, προστατεύσουμε ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από πόλεμο και βασανιστήρια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία δυνατότητα να ταξιδέψουν μόνιμα ως την Ευρώπη. Δεν έχουν θεωρήσεις, και αν θέλουν να φτάσουν ως εδώ, μπορούν ε, να το κάνουν αυτό μόνο παράνομα. Βεβαίως το σχόλιο του κυρίου Γιούνκερ ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί που χρήζουν προστασίας βάσει των νομικών υποχρεώσεων πρέπει να ε, φτάνουν με νόμιμες οδούς στην Ευρώπη. Αυτές οι νόμιμες οδοί δεν υπάρχουν, είναι σαφές. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Πριν από λίγο καιρό οι Πολωνοί χρησιμοποίησαν αυτές τις νόμιμες οδού μετανάστευση για να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ κύριε Κόμε. Ε, ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένη που το δικαστήριο ε, αποσαφήνισε τα πράγματα. Και πραγματικά θέλω και περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει οι χώρες που ε, αντέκρουσαν την απόφαση για την μετεγκατάσταση του Συμβουλίου να έρθουν αντιμέτωπες με τις ευθύνες τους. Όχι απλώς να δεχτούν την ποσόστοση ανθρώπων που τους αναλογεί, γιατί ακόμη υπάρχουν ε, μετανάστες που θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν, αλλά να ε, τους επιβληθούν κυρώσεις. Είμαι από την Πορτογαλία, θα το ξαναπώ. Μια χώρα που απειλήθηκε με κυρώσει από τα διευθυντικά ταμεία γιατί δεν ακολουθούσαμε κατά μονάδες ε, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Και δεν παραβιάσαμε για κανένα νόμο ούτε του διεθνούς δικαίου ούτε του ευρωπαϊκού. Όλα αυτά δεν ήταν ευρωπαϊκές συνθήκε αλλά και κυβερνητικές συμφωνίες και αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν κάποια κύρωση, κάποια ποινή να υπάρξει αν οι χώρε ε, που λέγαμε δεν, είναι, δεν εκπληρώνουν τις, υποχρεώσεις τους βάσει τη απόφαση του δικαστηρίου κιόλα. Ήθελα να ζητήσω από τους προσκεκλημένους μας από την Επιτροπή να μας πούν τι συμβαίνει με τις εισόδους στη Βουλγαρία. Από Τουρκία προς Βουλγαρία δηλαδή. Έχουμε στοιχεία και το έχουμε δει αυτό. Σε μια χώρα μειώνεται ο αριθμός, αυξάνεται σε άλλη. Μα ενδιαφέρει αν δήλωση με την Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, κατά την αντίληψή σα, λειτουργεί ε, σε όλα τα μέτωπα. Και ήθελα και να μου πείτε, γιατί μου είπατε τι γίνεται με τους ασυνόδευτούς ανηλίκους, και την περίπτωσή του στην Ιταλία και την Ελλάδα και την παρουσίασετε σαν να έχει όντως βελτιωθεί. Πολλέ από τι δυσκολίε που είχαμε είχαν να κάνουν με την έλλειψη δυνατοτήτων, την έλλειψη δικαστικών λειτουργών, εισαγγελέων να μπορούν να παρακολουθήσουν το τι συνέβη. Και αυτό που έγινε με του ανηλίκου είναι ότι εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, εξατμίστηκαν. Δεν μας νοιάζει αν κατέληξαν στα χέρια ε, εγκληματιών, δικτύων οργανωμένου εγκλήματο, Υπάρχει καμιά παρακολούθηση του όλου θέματο από τα κάτι μέλη. Έχουμε ακούσει να συμβαίνει άλλο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω για την Ιταλία ειδικά, αλλά και επίση λέτε ότι πιέζεται τι χώρε να τηρήσουν τι υποχρεώσει αλληλεγγύη που έχουν αναλάβει βάσει τη συμφωνία με την κατάσταση. Πρόσφατα είχαμε στοιχεία ότι κάποιε μεγαλύτερε χώρε που είχαν πολύ περισσότερε δυνατότητε να δεχτούν ανθρώπου από τη μετεγκατάσταση, το σύστημα μετεγκατάσταση από την Ιταλία και την Ελλάδα δεν απήχαν πολλοί από τους στόχους τους. Μια τέτοια χώρα ήταν η Ισπανία. Τι γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσει χώρες όπως η Ισπανία να παραμείνει πιστή σε αυτές τις υποχρεώσεις της. Και τι γίνεται με τις χώρες όπως η δική μου, η Πορτογαλία, που τα προβλήματα δεν είναι ότι εξωσυγνωρίζω το κατά πόσο είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε ανθρώπους από κατάσταση, αλλά ότι όταν φτάνουν οι μετεγκατεστημένοι, επειδή έχουν μείνει πολύ καιρό στην Ελλάδα ή αλλού, κανονίζουν για να πάνε σε δεύτερη φάση σε άλλη χώρα. Περίπου το 50% λένε τα στοιχεία. Οι μετεγκατεστημένοι στην Πορτογαλία τραπετεύουν, ξεφεύγουν, πηγαίνουν αλλού. Υπάρχει καμιά προσπάθεια να γίνει με την κατάσταση των ανθρώπων εκεί που θα έπρεπε να μετακατασταθούν αρχικά. Και τέλος η Λιβύη. Και θα το συνδυάσω με αυτό που είπε και τη Σίπελ μόλις τώρα. Εάν δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς οδοί, δεν εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Βάσει του διεθνού δικαίου έναντι των προσφύγων, όλος ιδιαίτερος. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν έγινε καμιά απόπειρα για μετεγκατάσταση ανθρώπων που βρέθηκαν στη Λιβύη και έχουν οριστεί ως πρόσφυγες. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, η υπατερμοστία του δεν έχει κάνει εκεί βάση για να δράσει στη Λιβύη. Δεν έχουν κανένα, καμιά δομή. Ίσως να έχουν κανένα δυο ανθρώπους, αλλά προφανώ δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, αλλά δεν είναι δική του εντολή να εντοπίζει του ε, πρόσφυγε. Είναι απλώ ε, να αναλαμβάνει τη σωματική του μεταφορά, να του διοργανώνει. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν ακριβώ στη Λιβύη. Με ανησυχεί πάρα πολύ διότι προ στιγμή στη Λιβύη με την έλλειψη κυβέρνηση ή τέλο πάντων τη κακή κυβέρνηση που επικρατεί ή την τριπλή κυβέρνηση που έχουν εκεί πέρα Πολύ φοβούμε ότι χρηματοδοτούμε την πλέον φρικαλέα μορφή ε, κράτηση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και βασανιστήριο. Κύριε Γιούρεκ, δευτερολογία, ερώτηση, επερώτηση. Ευχαριστώ. Ε, σε σχέση με όσα είπε ε, όχι μόνο η κυρία Γκόμες, αλλά και σε προηγούμενες παρεμβάσεις. Τα παιδιά είναι θύματα. Θύματα της παράνομης μετανάστευσης, της της μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το θέμα είναι λοιπόν τι υποστηρίζουν και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν δεν ήθελα τώρα να επιδείξω φιλική διάθεση προς την κυρία Κοντρίτσκα που είναι Πολωνή, αυτό που είπε για τους Πολωνούς και τους Ούγκρους που φεύγουν από τις χώρες τους ήταν άπρεπο και εσφαλμένο. Μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Όντως, Δεκάδες χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ των Ηνωμένων Βασιλείων. Μιλάμε όμως για στρατιώτες που προδόθηκαν. Πολλοί είναι οι Ουγγροί που έφυγαν από την Ουγγαρία το 1956. Είναι άνθρωποι όμως που περασπίστηκαν την Ευρώπη και τους πρόδωσε η Ευρώπη. Πολλοί έφυγαν ε, λόγω του, ε, της κατάστασης έκταξης ανάγκης και ε, του στρατιωτικοποιημένου κράτους. Και τώρα μιλάμε για, ανθρώπου, για κράτη που θέλουν να κάνουν λιγότερες δαπάνες στον τομέα της άμυνας και το ενεργητικό. Ε, η Ευρώπη τους πρόδωσε. Ε, για, μιλάμε για χώρες που προκάλεσαν φρίκη και πόλεμο. Ε, η κυρία Γκόμες ε, εργάζεται μαζί μου στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Πρέπει να καταλαβαίνει το πόσο διαφορετικά πράγματα είναι αυτά που ε, διέπουν την ε, κατάσταση ειρήνη που ζούμε στην Ευρώπη και τις εγκληματικές οργανώσεις της λαθρομετανάστευση. Βεβαίω πρέπει να ε, βοηθήσουμε του πρόσφυγε πολέμου, πρόσφυγε, αλλά εδώ μιλάμε για μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω έχει καθημερινά συνεργασία με τη Frontex και πολλοί από εμά μπορούμε να γίνουμε καθημερινά μάρτυρες του τι συμβαίνει. Αν πάμε στην Αμερικανική πρεσβεία, θα δείτε πώ πάνε οι άνθρωποι να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Έποτε τους νόμους, ακολουθεί μια διαδικασία για να πάνε. Άλλο είναι ένα καταβλισμός προσφύγων με κάποιον που θέλει να είναι πολιτικό πρόσφυγα. Εάν κάποιο μπορεί να αποδείξει ότι διώχθη, φυσικά είναι υποχρεώσει κάθε πολιτισμένη χώρα, να τον αναλάβει. Αλλά εδώ τι λέμε. Ε, πραγματικά θέλουμε να έχουμε και άλλε τέτοιες τραγικέ περιπτώσει και καταστροφές όπως αυτές αυτών των παιδιών που είδαμε, ε, το ξέρουμε πολύ καλά, ε, τα συζητάμε στο κοινοβούλιο. Ποιοι είναι πίσω από αυτά, ποιες είναι αυτές οι μαφίες, αυτοί οι λαθρέμποροι που τα προκαλούν όλα αυτά. Μιλάμε για τεράστια συμφέροντα, είναι πολύ το χρήμα πίσω από αυτές τις ε, ιστορίες. Δεν μπορούμε λοιπόν εμεί να πάρουμε την ευθύνη των εκτελεστικών εξουσιών των διαφορών χωρών που προέβλεψαν τέτοιε πολιτικέ. Απλώς λοιπόν θα σας προειδοποιήσω, θα σας προειδοποιήσω ξανά. Είναι δύσκολο να ε, κάνει κανείς έφεση κατά των αναδικαστικών αποφάσεων, αλλά μας δίνουν ε, αφορμή να σκεφτούμε το κράτος δικαίου. Επιβάλλουν μια νομολογία, αλλά δεν μας απε, απαλλάσσουν από κάθε πολιτική ευθύνη. Είμαστε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωση και πρέπει να συνεργαστούμε προς το σωστό σκοπό. Ευχαριστώ, Σόφη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, πέντε δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που ακούω τον κύριο Γιούρεκ, πάντοτε μιλάει για τις χριστιανικές αξίες. Αλλά δεν το βλέπω ποτέ να απεικονίζεται στα λόγια σας. Ποτέ δεν έχω ακούσει κουβέντα, καμιά κουβέντα για τη διαδεοδορία, για καλό γείτονα, για προσφορά καταφυγείου σε αυτούς που το χρειάζονται. Καμιά μέρα ίσως να μου το εξηγήσατε. Ε, τι εννοείτε με αυτές τις αξίες. Ευχαριστούμε κυρία Μετσόλα. Ρομπέρτα. Α, η Ανδρέα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να επαναλάβω αυτό που όλοι είπατε. Τα λόγια του Πρωθυπουργού Όρμπαν για την δικαστική απόφαση. Ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία θα αποδεχθεί την απόφαση του δικαστηρίου. Μπορώ να σας πω ακριβώς και τα λόγια του. Μια απόφαση δικαστηρίου μόλις εκδόθηκε. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να παραμείνουμε στη θέση αυτή. Η Ουγγαρία είναι ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, οι εξουσίες ορίζονται βάσει των ιδρυτικών συνθήκων. Οι συνθήκες πρέπει να γίνουν σεβαστές, τη απόφαση του δικαστηρίου. Και βάσει των ε, της δήλωσης του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας και της Πολωνίας πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε και εμείς τη δικαστική απόφαση προκειμένου να μην πλήξουμε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει σεβασμός για το κάτω δικαίου που είναι ένα από τα, μια από τις θεμελιώδεις αξίες της. Αυτό ήταν το παράθεμα. Να είστε βέβαιοι ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει πλήρως και σέβεται τη δικαστική αυτή απόφαση. Όμω δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να, λέει η κυρία Γκόμε που να τιμωρηθεί η Ουγγαρία ή οι άλλε χώρε. Διότι κάποιε χώρε δεν λένε τίποτα, αλλά δεν κάνουν καμιά κατάσταση. Είναι πολύ πιο εύκολο να μην ακολουθεί κανείς τους κανόνες και να μην λέει και τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε. Κάθε χώρα να κάνει αυτό που της αναλογεί. Όπως θεωρεί ότι αυτό είναι το δέον και το καλύτερο. Ευχαριστώ. Να... Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Κύριε Φερβέν. Uh, Ο κύριος Φερβέη. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, θα σχολιάσω τα, τις διάφορες παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Καταρχάς, και θέλω να είμαι σαφής. Η κυρία Ίνφελτ είπε ότι δεν άκουσε τίποτα για τον κόσμο. Μπορεί να εκφραζόμαστε διαφορετικά, αλλά αν εκφράσω τις ανησυχίες μου για τις συνθήκες στα νησιά και όταν μιλώ με αυτούς τους όρους, τους ανθρώπους σκέφτομαι. Ε, με ρωτήσατε για τις συνθήκες υποδοχής στην Τουρκία, πόσα παιδιά πάνε σχολείο. Οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση, την αντίστοιχη, νομίζω μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Να σας πω το εξής, δεν μπορώ να εγγυηθώ και δεν θα εγγυηθώ ότι κάθε παιδί από τη Συρία που βρίσκεται στην Τουρκία πράγματι πηγαίνει σχολείο και ότι όλοι ε, ε, γίνονται αντικείμενο τέλειας φροντίδας. Αυτό που σίγουρα μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλά περισσότερα παιδιά πάνε στο σχολείο από ό,τι πριν και πολλοί περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι πριν έχουν πρόσβαση σε ε, καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας, περίθαλψης, λοιπά. Αλλά τις λεπτομέρειες θα παρουσιάσουν οι συνάδελφοι από την αντίστοιχη και αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Με ρωτήσατε αν εξετάσαμε το κατακεφαλήν κόστος για τις επιστροφές και αν είναι χρήματα καλά δαπανημένα, money well spent. Εγώ είμαι οικονομολόγος, ξέρετε, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν σας λέω ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να εξετάζει κανείς το πρόβλημα το προσφυγικό. Σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι θα υπάρξουν που θέλουν να δουν και τα οικονομικά του θέματος της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τα, αν το πράξουν τα μαθηματικά μετατρέπονται σε αριθμητική απλή. Είναι πολύ πιο δαπανηρό να φροντίσουμε ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σαφέστατο και είναι απλά μαθηματικά, αλλά επιμένω ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος να εξετάζει κανείς το ζήτημα, αλλά αφού το αναφέρεται οφείλω και εγώ να το σχολιάσω και να το πω. Τώρα, για το κόσμο στα νησιά για το άγχος, για το στρες και το καθεξής. Και εδώ ακριβώς έγκυται η ανησυχία μου. Δύο είναι τα στοιχεία του στρες και του άγχους. Υπάρχει στρες, πίεση και άγχος γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του γιατί πρέπει να περιμένει πάρα πολύ και αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι οι υφιστάμενες συνθήκες διαβίωσης. Νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί στα νησιά, στο νησί είναι το εξής έχουμε κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν είμαι ικανοποιημένο με τις υφιστάμενες συνθήκες επιτόπου στα νησιά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει υπερπληθυσμός. Μπορώ να σας πω για τις βελτιώσεις, την διοργάνωση, για τους έξτρα ανθρώπους, για τις υπηρεσίες εστίασης, για τους έξτρα γιατρούς που έχουν καταφτάσει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τη χωρητικότητά τους και αυτό δημιουργεί προβλήματα και είναι πραγματική ανησυχία. Τώρα, για το άλλο είδος ανησυχίας και άγχους, Υπάρχει βεβαίως το άγχος για τους ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορούν. Πράγματι, θα έλεγα όμως ότι αυτό το κομμάτι έχει μετριαστεί κάπως γιατί έχουν μειωθεί και τα περιστατικά ασφαλείας. Αυτό φαίνεται από τη μείωση των περιστατικών ασφαλείας, γιατί ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι αυτοί στα νησιά έχει μειωθεί δραματικά. Αυτή η ατέρμονη αναμονή που περιμένει κανείς το πρώτο του ραντεβού, περιμένει την πρώτη του συνέντευξη, αυτό είναι αυτό που δημιουργούσε πάρα πολύ ένταση και πολύ άγχος. Σίγουρα ε, ε, στρες έχουν και αυτοί που παίρνουν μια δεύτερη αρνητική απάντηση γιατί δεν θέλουν να επιστρέψουν. Αλλά το μη απαραίτητο άγχος του να πρέπει κανείς να περιμένει χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί και χωρίς να έχει καμία πληροφορία, νομίζω ότι ως προς αυτό το κομμάτι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Από εκεί και πέρα Κατά πόσο φοβάμαι αν έρθουν οι πρόσφυγες από την Τουρκία εδώ και ότι θα το χρησιμοποιήσει αυτό η τουρκική κυβέρνηση ως ε, ε, μάρκα για το ποντάρισμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κτλ. κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα να ανησυχώ εγώ ή όχι το αντίθετο και δεν νομίζω ότι έχει και καμία σημασία και ευτυχώς και δόξα τω Θεώ δεν είμαι εγώ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι πολιτικοί που αποφασίζουν το κατά πόσο κάποιος θα επιστρέψει ναι ή όχι. Το αποφασίζει αυτό ε, ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, ανεξάρτητες δικαστικές αρχές. Επομένως, Νιώθω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη με το γεγονός ότι μπορεί να ασκηθεί πολιτική πίεση, ενδεχομένως, αλλά δεν θα αλλάξει και τίποτα γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γι' αυτό. Τώρα, δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τα κράτη-μέλη. Και αν πρέπει να ασκήσω κριτική να... στα κράτη-μέλη θα το πράξω και νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνουμε και ασκούμε κριτική στα κράτη-μέλη. Σε κάθε περίπτωση θέλω όμως να πω τα εξή. Το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες τα νησιά σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την έλλειψη χρηματοδότησης. Δεν είναι δηλαδή ότι αν είχαμε δώσει περισσότερα λεφτά στα κρατημέλη θα είχαν βελτιώσει την κατάσταση. Υπάρχει επαρκή σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και κινητοποιούμε πόρους κτλ. Η ουσία του ζητήματος έγκυται στο ότι η χωρητικότητα δεν αρκεί. Ο χώρος δεν αρκεί. Ο χώρος δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Δεν φτάνουν οι εγκαταστάσεις για τον αριθμό των ατόμων που μένουν εκεί το έχω πει και προηγουμένως και επανειλημμένως αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο με την τοπική κοινότητα να υπάρξει συμφωνία για να έχουμε περισσότερους χώρους εγκαταστάσεων. Και αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Και αυτό ήταν ένα από τους βασικούς λόγους που πήγα και την προηγούμενη εβδομάδα στη Λέσβο για να συζητήσω ξανά και ξανά για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε ως προς αυτό. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τα κρατη για άλλα, αλλά όχι γι' αυτό κατά τη γνώμη μου. Για τη μετεγκατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει ορισμένες δράσεις στο θέμα μετεγκατάστασης, αλλά θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Δεν είναι απολύτως σωστό και ορθό να επανέρχεται κανείς στο ζήτημα ότι είναι κρίμα ότι 66.000 δεν μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα, γιατί δεν υπήρξαν, δεν υπάρχουν 66.000 Σύριοι που θα μπορούσαν να είχαν μετεγκατασταθεί και δεν μετεγκαταστάθηκαν. Δεν είναι εκεί παρόντες, δεν υπάρχουν 66.000 Σύριοι. Άρα αφού δεν υπάρχουν δεν μπορεί κανείς να τους μετεγκαταστήσει. Πρέπει τώρα να προχωρήσω λίγο γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει στο ζήτημα και αν το κατάλαβα καλά. Οι 1920 επιστροφές πώς συνδέονται, στην Τουρκία πώς συνδέονται με την Ιταλία. Η απάντηση είναι δεν συνδέονται, δεν έχουμε επιστροφές από την Ιταλία στο βαθμό που γνωρίζω εγώ. Και μετά, για το πώς ε, εξηγούμε την αύξηση των αφήξεων στα νησιά. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ότι υπάρχει μια εποχικότητα σε αυτή τη τάση. Πέρσι τον Αύγουστο, για παράδειγμα, είχαμε 110 αφήξεις την ημέρα και φέτος 117. Λίγο περισσότερες, αλλά όχι δραματικά ψηλότερες. Το Σεπτέμβριο Είχαμε πολλές αφήξεις. Κατά μέσο όρο 460 την ημέρα και πέρσι 100 την ημέρα το Σεπτέμβριο. Αλλά και πάλι αυτό είναι, είναι λίγο σε σχέση με ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν. Προσπαθώ, Προσφανώς προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε κατά πόσο υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν έχουμε τέτοιου είδου ενδείξει. Δεν έχουμε σαφείς εξηγήσει για τις ε, ε, παρεμποδίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει ακολουθούνται οι συνήθεις ροέ. Ε, ένα μέλος της Επιτροπής σας αναφέρθηκε σε ένα σχόλιο που είχα κάνει για τον αριθμό των θανάτων και των εξαφανισμένων στο Αιγαίο και λογικό είχε πολύ το δικαίωμα το μέλος της Επιτροπής να αναφερθεί σε κάθε τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση εγώ έχω να πω ότι δεν το βλέπω ως αναλογία και ως λόγο και ως ποσοστό παρόλο που είμαι οικονομολόγος. Το σημαντικό για μένα δεν είναι ε, ε, ε, τα νούμερα. Είτε 1.100 πεθαίνουν είτε 100, το ίδιο σημαντικό είναι. Για την Ουγγαρία δεν έχω σαφή εικόνα. Για τη Βουλγαρία με συγχωρείτε για το τι συμβαίνει. Εξετάζοντας τα νούμερα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση. Ίσως υπάρχει μια κάποια αύξηση και εγώ διαβάζω τις ίδιες εκθέσεις, τις ίδιες αναφορές ότι ο κόσμος δοκιμάζει άλλες μεταναστευτικές και προσφυγικές οδούς. Μοιραία θα συμβεί κάτι ε, τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι μιλώντας ε, με βάση τα νούμερα είναι πολύ περιορισμένα και χαμηλά ακόμα, μικρά. Και ίσως το τελευταίο που θα ήθελα να πω ε, έχει να κάνει με τη Λιβύη και τις νόμιμες οδούς διέλευσης. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για τη Λιβύη, δεν είμαι έτοιμος να σχολιάσω γι' αυτό, δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Η τελευταία μου παρατηρήση έχει να κάνει με τη σημασία των νομίμων οδών ε, διέλευσης. Κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να έχουμε καταστάσεις όπου εξαιρετικά ευάλωτοι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τους είτε για να διασχίσουν τη Μεσόγειο είτε για να διασχίσουν το Αιγαίο. Επομένως, ακόμα και αν διαφωνείτε με οτιδήποτε άλλο έχω να πω, σίγουρα σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι και ο τρόπος να το πετύχουμε είναι Αντί να έχουμε τις παράνομες οδούς ε, διέλευσης, να προσπαθήσουμε να νομιμοποιήσουμε κάποιες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίλσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τη συνέχεια που θα δοθεί στην απόφαση, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έστειλε επιστολή στους Υπουργούς Δικαιοσύνης των χωρών μελών, περιμένουν βέβαια την απάντησή τους, ενθαρρύνοντάς τους να συμμορφωθούν με την απόφαση. Όσο τώρα το πώς πιέσαμε τις χώρες μέλη προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα και τα λοιπά, το έργο γίνεται και πολιτικά, αλλά και συνεργαζόμαστε στενά με τις χώρες μέλη. Οι αξιωματούχοι στην Αθήνα και την Ρώμη είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Βλέπουμε κάποια πρόοδο. Ξέρω ότι υπάρχουν λόγοι για απογοήτευση, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα, πολλά που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη έκθεσή μας, τώρα δεν προκύπτουν. Όλοι έχουν πει ότι πρέπει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση όμως δεν είναι τόσο ζωβερή. Πρόοδος έχει γίνει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απολύτως ό,τι αφορά την Ελλάδα. Δεύτερο στοιχείο, για κάποια κάτι μέλη απλώς δεν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο κύριος Φερβέη, ε, μερικοί απλώς δεν υπήρχαν για να μετεγκατασταθούν. Επίσης, για την, ε, με την κατάσταση γιατί να μην είναι και νομικός δεσμευτικό, ίσως. Κάποια κάτι μέλη, τα περισσότερα, έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όπως είπα, σε σχέση με όσα είχαν αποφασιστεί το 2015, ε, θα πρέπει να το κάνουν όλοι για να υπάρξει ισορροπία. Σε ό,τι αφορά τι δεύτερε μετακινήσει ανθρώπων που έχουν μετακατασταθεί, των μετεγκατεστημένων, αυτό ήταν πρόβλημα για ορισμένα κράτη-μέλη. Η συνολική όμω εικόνα ε, δείχνει ότι είναι η εξαίρεση. Από τα διδάγματα που αντλήσαμε από τα προγράμματα αυτά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δύο πράγματα είναι σημαντικά ε, τη στιγμή που κάποιο φτάνει στο κράτο με την κατάσταση, θα πρέπει να υπάρχουν καλέ εγκαταστάσει υποδοχή. Όχι μετά από μια εβδομάδα, τη στιγμή που κάποιο βγαίνει από αεροπλάνο. Ε, στην ουσία. Αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά ε, το, για το αν οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να πάνε αλλού μετά ή όχι. Επίση, θα πρέπει οι κανόνε απλώ να εφαρμόζονται. Δηλαδή, όταν κάποιο όντω ε, μετακινείται σε δεύτερο κράτο, θα πρέπει να ισχύει το Λουβουβλίνο, να πηγαίνει στο κράτο με κατάσταση, δηλαδή ξαναπίσω. Αυτό είναι σημαντικό τα κάτι μελη να το λένε στου πρόσφυγε. Δεν μπορούν να επιλέγουν ελεύθερο ό,τι του αρέσει. Υπάρχει κάποιο κράτο μέλο που είναι υπεύθυνο για τον καθένα. Όσο για τους ανηλίκους, οι αριθμοί ε, για την Ελλάδα, όπως λέγει και η έκθεση, έχουν μετακαταστήσει 420 από τους 586 ε, ανασυνόδευτους ανελίκους. Ο αριθμός αυτός ίσως είναι κάπως μεγαλύτερο σήμερα γιατί ήδη έχει περάσει 15 φήμερα από το που τα καταγράψαμε. Στην Ιταλία είμαστε στους 31 ε, συνόδευτους ανελίκους σε αντικατάσταση. Μικρό φαίνεται ο αριθμό, αλλά εάν ε, συγκριθεί με το μηδενικό αριθμό πριν από τέσσερι μήνε, τουλάχιστον δείχνει ότι κάτι έγινε. Και υπήρξε ε, συμμόρφωση με τι συστάσει που κάναμε, η διαδικασία έρχεται να λειτουργεί και υπάρχουν και κάποιε δεσμεύσει ε, που εφαρμόζονται του τελευταίου τουλάχιστον τέσσερι μήνε. Είναι χαμηλό αριθμό, αλλά ελπίζουμε ότι η πρόοδο θα συνεχιστεί. για το ποιο εμπίπτει το, εντός αυτών των 5-6 που πρέπει ακόμη να ε, μετεγκατασταθούν είναι άνθρωποι που μόλι έχουν φτάσει. Εκτιμούμε ότι οι περισσότεροι είναι στην Ιταλία. Λόγω των καθυστερήσεων που είδαμε στην Ιταλία στην καταγραφή αυτών των ε, ανθρώπων με την κατάσταση καθυστερεί. Και θα πάνε όλα καλά, ελπίζουμε, στη συνέχεια, προκειμένου ο αριθμό αυτό να συμπληρωθεί. Όσον αφορά τώρα τι περιπτώσει που δεν υπάρχει συνέχεια. Οι εκτιμήσεις μας είναι εκτιμήσεις, γιατί η κατάσταση αλλάζει και από μέρα σε μέρα. Για την επανεκατάσταση τα είπε και ο κύριος Φερβέ, πάντα ήταν σαφής η Επιτροπή ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και να αποφύγουμε την παράτυπη μετανάστευση. Έχουμε πει τι θα ήταν η φιλοδοξία μας για κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει ένας νόμιμος τρόπος για αυτή τη μετανάστευση. Για τη Λιβύη, το θέμα νομίζω έχει να κάνει περισσότερα με τα Ηνωμένα Έθνη, που αγωνίζονται να έχουν προστασία για το δικό τους το προσωπικό πρώτα απ' όλα. Αν το είχαν αυτό, θα μπορούσαν να είναι περισσότερο παρόντες στη Λιβύη και να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους. Από πλευρά της Επιτροπής, γι' αυτό προτείναμε στις χώρες μέλη να συμπεριλάβουν τις περιπτώσεις αυτές. Σήμερα δεν γίνεται. Αλλά αν οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, θα ήταν θετικό. Σίγουρα είπα την αρμοστία του ΟΗΕ το προχωράει. Συγγνώμη αν δεν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά εντάξει, πολύ σύντομα εσείς. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ όσον αφορά τη διευκόλυνση, τα 3 δηλαδή δισεκατομμύρια, που είναι χρήματα για τους πρόσφυγες, όχι για την Τουρκία. Μέχρι τώρα έχουμε δεσμευτεί για τα 2,9 και περιμένουμε ακόμα για το 1,7. Πάντως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε τα 3 δισεκατομμύρια. Έχουμε χρηματοδοτεί 49 διαφορετικά προγράμματα μέχρι τώρα με κυβερνητικέ υπηρεσίες, Ινστιτούτα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις προκειμένου να προσφέρουμε ανθρωπιστική και μη ανθρωπιστική αρρωγή στους πρόσφυγες. Παράδειγμα, έχουμε τρεις συμβάσεις με τις τουρκικές αρχές. Ένα θέμα είναι η εκπαίδευση για 500.000 παιδιά προκειμένου να πάνε στο σχολείο στην Τουρκία. Και χρηματοδοτούμε και πρωτογενή και δευτερογενή περίθαλψη. Όπως επίσης και την οικοδόμηση 200 κατοικιών. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα είναι έτοιμη το Μάρτιο. ήταν έτοιμη το Μάρτιο. Υπάρχουν πληροφορίες για τη δομή, για το πώς λειτουργεί η διευκόλυνση αυτή. Διακόπτη Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έπρεπε να είχαμε τελειώσει πριν από 10 λεπτά. Τελευταία σας πρόταση. Είναι υπεύθυνη μια steering committee για τη διευκόλυνση αυτή προς την Τουρκία, η οποία θα συνεδρίασει πάλι τον Αύριο. Όχι, λυπάμαι. Σίγουρα πολλές ε, θα ήταν οι συζητήσεις στο μέλλον. Το επόμενο θέμα έχει αναβληθεί για τις 12 Οκτωβρίου που θα ψηφίσουμε. Μην το ξεχνάτε. Μάλλον για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στο Στρασβούργο θα συνεδριάσουμε και πάλι 5 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ.